Uh, uh, λοιπόν, να σας καλωσορίσω καταρχήν όλους. Εγώ θα πρέπει να ξεκινήσω αυτή την ε, ακρόαση που είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί θα μας δώσει σήμερα την δυνατότητα να εμβαθύνουμε ε, στην πρόταση της Κομισιόν, την πρόταση οδηγίας ε, σε σχέση με την καταπολέμηση της κατάχρησης και της, ε, των παιδιών και την παιδική πορνογραφία και όπως ξέρετε αυτή θα αντικαταστήσει την απόφαση πλαίσιο του 2004. Εγώ θα πω μόνο δύο λόγια γιατί στόχος ε, μιας ακρόασης είναι ακριβώς να ακούσουμε ε, τους εμπειρογνώμονες. Θα είναι λοιπόν για μας σημαντικό να καταγράψουμε με μεγάλη προσοχή ε, όλες τις συμβολές των προσκεκλημένων μας. Νομίζω πως είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε τρεις επιτυχές αυτής της οδηγίας που κατά την άποψή μου θέτει πολύ συγκεκριμένες προτεραιότητες και είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη. Καταρχήν, να καταστήσει πιο αποτελεσματικές τις κυρώσεις για όσους διαπράττουν τέτοιου είδους εγκλήματα. Μια άλλη πτυχή που μου είναι ιδιαίτερα προσφυλής είναι αυτή μιας καλύτερης προστασίας και βοήθειας στα θύματα βίας και κατάχρησης. Και έπειτα είναι σημαντική μια στρατηγική μακρόπνοη που στόχο έχει την πρόληψη όχι μόνο από νομοθετική άποψη, αλλά και από ενημερωτική άποψη, επικοινωνική άποψη και κοινωνική άποψη. Αυτή η πρόταση οδηγίας προκύπτει από μια σαφή ε, υπόδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μάλιστα πρόσφατα Το 2009 μόλις ζήτησε από την Επιτροπή μια αναθεώρηση της απόφασης πλαισίου του 2004. Αυτή η πρόταση σίγουρα περιλαμβάνει εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία. Να αναφέρω μερικά και κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντική η εισαγωγή των επιβαρυντικών στοιχείων. Είναι επίσης πολύ σημαντικός ο στόχος της ε, αποσαφήνισης του τι εννοούμε όταν μιλάμε για σεξουαλικό τουρισμό και με ποιο τρόπο θα πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτό το όλο ένα και αυξανόμενο φαινόμενο. Στόχος η καταπολέμηση επίσης της παιδικής πορνογραφίας online και Ακριβώς για αυτό το θέμα έχει ξεκινήσει μια ευρύτατη συζήτηση που θα είναι σημαντικό να ε, ε, διευκρινιστεί και εδώ κατά τη διάρκεια του ακρόασης. Άλλη σημαντική ε, πρωτοβουλία είναι η, ο ορισμός του, του εγκλήματος online του grooming όπως λέγεται Δηλαδή οι ανήλικοι ε, έχουν να αντιμετωπίσουν διπλή διάκριση. Δηλαδή καταρχήν τους ασκείται βία, ή ε, γίνεται κατάχρηση των αυτούς και έπειτα κατά κάποιο τρόπο πέφτουν θύματα των ε, ΜΜΕ που παραβιάζουν τη δική, ιδιωτική τους ε, ζωή, πέφτουν θύματα και δικαστικών διαδικασιών που δεν ε, λαμβάνουν υπόψη την ιδιαίτερη, την ιδιαίτερα ευάλωτο χαρακτήρα ενός ανηλίκου. Γι' αυτό και νομίζω ότι έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Εδώ λοιπόν ολοκληρώνω την παρέμβασή μου και θα ζητήσω από τους ομιλητές να τηρήσουν το χρόνο τους. Θα είμαι αυστηρή σε αυτό και θα δώσω αμέσω το λόγο στον κύριο Κάμερβερτ που αντιπροσωπεύει την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και που είναι αρμόδιο για τη σύνταξη μιας ε, γνωμοδότησης για αυτό το θέμα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μπορώ να είμαι εδώ σήμερα ως εισηγήτρια σε αυτή την ακρόαση για, από την Επιτροπή Πολιτισμού ως συντάκτρια της έκθεσης και της νομοδότησής μου για να σας αναφέρω ποιες είναι οι σκέψεις μου. Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου πριν μπω στα βασικά σημεία της ε, γνωμοδότησής μου να κάνω κάποιες αρχικές παρατηρήσεις. Ε, πολύ γρήγορα έμαθα ότι πρέπει πάντα να λέμε ή να τονίζουμε ότι η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών και των εφήβων ε, είτε και η παρουσίασή της είτε στον πραγματικό είτε στον ε, ψηφιακό κόσμο αποτελεί ένα από τα, βασικό, από τα απεχθέστερα εγκλήματα που μπορεί να ε, κάνει κάποιος. Πρέπει να διώκονται οι δράστες και να πηγαίνουν βρίσκονται ενώπιον του δικαστηρίου. Επίσης, η χρήση αυτών των ε, ε, αποδεικτικών στοιχείων των ε, φωτογραφιών από σεξουαλική κακοποίηση παιδιών δεν καλύπτεται από την ελευθερία πληροφόρηση και ενημέρωση. Επίση, στον πραγματικό κόσμο, όπω και στον ψηφιακό κόσμο, υπάρχει εγκληματικότητα. Οπότε πρέπει να αντιμετωπιστούν και στους δύο κόσμους και να, τις, να προσπαθήσουμε να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να γίνει αυτό. Το ίντερνετ δεν είναι ελεύθερος χώρος, είναι ένας χώρος στον οποίο πρέπει να ισχύουν οι κανόνες που ισχύουν και στον πραγματικό κόσμο. Πρέπει να μιλούμε για ε, ελέγχους, ε, για ε, μέσω των οποίων μπορεί η Κομισιόν να αντιμετωπίσει την σεξουαλική εκμετάλλευση, την κακοποίηση και πρέπει να προωθήσουμε την δίωξη των ατόμων που κακοποιούν σεξουαλικά άτομα κατά των 18 ετών ανηλίκους. Πρέπει να δημιουργήσουμε νέου ε, ε, ε, τρόπου για να το αντιμετωπίσουμε αυτά, γιατί οι νέε τεχνολογίε οξύνουν το πρόβλημα. Οπότε πρέπει να βρούμε ανάλογα και εμεί ανάλογε λύσει. Πρέπει να καθορίσουμε συγκεκριμένε ποινέ, πρέπει να υπάρξουν ποινικέ καθήρξει. Όλα αυτά πρέπει να είναι στη διάθεση της κοινωνία και εδώ η εποπτεία θα πρέπει να γίνει κυρίως στις τηλεπικοινωνίες συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής εποπτείας. Υποπτία ε, των ε, οικονομικών στοιχείων ή των ε, λογαριασμών των δραστών. Επίσης, τέτοια, αυτή η εποπτεία αυτη η εποπτεια μπορει να μπορεί να βοηθήσει ώστε να αντιμετωπιστούν τέτοια κρούσματα. Επίσης έχουμε το θέμα της ε, ε, αποθήκευσης των ε, δεδομένων όπως ισχύει τώρα στην Γερμανία, τα δεδομένα αυτά σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να μπορούν να τίθενται στην διαθεσιμότητα του δικαστηρίου. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε όλα αυτά να τα πετύχουμε με την οδηγία. Νομίζω ότι σε πολλά θέματα η οδηγία δεν φτάνει εκεί που πρέπει και σε πολλά άλλα σημεία ξεπερνά τους στόχους. Επίσης, στην Επιτροπή Πολιτισμού το συζητήσαμε ε, ότι πρέπει να ε, επενδύσουμε στην πρόληψη. Ε, υπάρχουν λοιπόν αρκετέ προτάσει από την Επιτροπή Πολιτισμού όπου μπορεί η οδηγία να ενισχυθεί. Επίσης, ένα βασικό κομμάτι είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα, μια εκπαίδευση ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες των ΜΜΕ δεν μιλούμε δηλαδή για την ε, τεχνογνωσία και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, αλλά την ε, ενημέρωση, την ανταλλαγή γνώσεων για το πώς μπορεί δηλαδή κανείς να διαχειρίζεται το ίντερνετ, τι πρέπει να αξιολογεί, ποιες πληροφορίες πρέπει να αποφεύγει. Οι νέοι και τα παιδιά πρέπει από νωρί να μαθαίνουν ε, να διαχειρίζονται το ίντερνετ, να γνωρίζουν ποιε είναι οι δυνατότητες που τους δίνει και ποιοι είναι οι κίνδυνοι και βεβαίω μετά να μπορούν κριτικά από μόνοι του να αποφασίσουν ποιο, τι ακριβώ θέλουν να κάνουν στο ίντερνετ, ποιε πληροφορίε θέλουν να δώσουν και ποιε όχι. Πρέπει λοιπόν να εξηγήσουμε στα παιδιά μα πώ ακριβώ μπορούν να, να ε, διαχειριστούν τον κόσμο του ίντερνετ. Να τους δώσουμε δηλαδή συγκεκριμένους τρόπους πώς μπορούν να ξεχωρίσουν το καλό και το κακό από μόνα τους. Δεν μπορούμε να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου το τέλος ε, όπου κάθε ένας που βοηθάει ένα παιδάκι στην παιδική χαρά επειδή έπεσε να θεωρείται κατευθείαν ύποπτο για σεξουαλική κακοποίηση. Πρέπει να υπάρχει ε, μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ εμπιστοσύνη ε, και ε, ποινικοποίηση. Επίσης, η σεξουαλική εκπαίδευση θα πρέπει να ενισχυθεί στα, στα σχολεία. Ε, μιλούμε για παλαιότερες ε, γενιές οι οποίες ε, δεν έχουν μεγάλη σχέση με όλο αυτό. Πολλοί γονείς ακόμη δεν ξέρουν τι ακριβώς κάνουν τα παιδιά τους στο ίντερνετ, τι σελίδες βλέπουν. Δεν μπορούν λοιπόν να απαντήσουν άμεσα. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν άμεση ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών. Πρέπει μονίμως να, ενημερώνονται τα στοιχεία αυτά, να βρούμε ποια είναι οι βέλτιστες πρακτικές, ποια είναι τα καλά παραδείγματα, ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε, να ενισχύσουμε την πρόληψη και να μάθει ο ένας από τον άλλον. Επίσης, η πρόταση για τη βελτίωση της συνεργασίας ε, αστυνομικών και ποινικών αρχών και των ε, παρόχων, ε, και των παρόχων ε, τηλεπικοινωνιών και ίντερνετ. Γιατί έτσι μέσω αυτών έρχονται σε σύνδεση, έρχονται σε επαφή τα παιδιά με τους πιθανούς ενδυνάμει ε, παρανόμους. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, συγκεκριμένα μέτρα ώστε να μπορέσουμε με τα βέλτιστες πρακτικές που υπάρχουν να τις χρησιμοποιήσουμε και να προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης, της ε, εκπόρνευσης ε, των ανηλίκων. Και αυτό πρέπει να γίνει ώστε το δυνατόν πιο γρήγορα. Επίσης, μπαίνω σε έναν τομέα όπου η Κομισιόν, νομίζω ξεπερνά τον στόχο για την διαγραφή των σελίδων με φωτογραφίες από κακοποίηση παιδιών και νέων. Η Κομισιόν μέσω αυτό, αυτού θέλω να, ε, θέλει να προβλέψει την απαγόρευση αυτών των σελίδων. Το συζητήσαμε και εμείς στην ε, Επιτροπή ε, Εκπαίδευσης αυτού και είπαμε ότι ε, θα πρέπει να γίνεται περισσότερο διαγραφή παρά ε, απαγόρευση αυτών των, ε, αυτών των παιδιών. Οι απαγορεύσεις δεν είναι κατάλληλο εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα κρούσματα. Δεν βοηθούμε τα παιδιά μας έτσι. Η απαγόρευση του ίντερνετ έχει δείξει και σε χώρες που το έχουν κάνει ότι δεν δεν βοηθά γιατί υπάρχουν πολλές σελίδες που σου δείχνουν πώς να ξεπεράσεις την απαγόρευση στο ίντερνετ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Πολλοί ε, ξεκινούν να δημιουργήσουν μία ε, δομή ε, ελεγκτική Βεβαίω δεν πρέπει να τα βάλουμε όλα στο ίδιο σακί, δηλαδή δεν μπορούμε να, απαγορε... να... να απαγορεύσουμε τα πάντα. Υπάρχουν και τομεί που πλήττονται μεν αλλά δεν είναι υπεύθυνοι, όπω α πούμε ο τομέα τη ε, μουσική. Επίσης το υλικό που μπορεί να ποινικοποιηθεί και μπορεί να, να τύχει η κατάκριση σε αν βρεθεί σε λαθασμένα χέρια. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Οι απαγορεύσεις δεν νομίζω ότι μπορούν να οδηγήσουν σε αυτό το, στο αποτέλεσμα που θέλουμε εμείς. Θέλουμε να μπορέσουμε να έχουμε άμεση διαγραφή όλων αυτών των σελίδων και του περιεχομένου που περιλαμβάνουν, ώστε να μπορέσουμε να εποπτεύσουμε καλύτερα, να διαγράφονται άμεσα οι ε, σελίδες αυτές. Και μετά από μία έρευνα είδαμε ότι το 98% ε, διαγράφεται, των σελίδων αυτών διαγράφεται μέσα σε μία εβδομάδα όταν βρεθεί και ε, ποινικοποιηθεί. Αυτό όμως θα πρέπει να το καθορίσουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν θα μπορέσουμε τώρα να φτάσουμε σε ένα συμβιβασμό, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να το αφήσουμε αυτό στο κράτη-μέλη. Ίσως αν θεωρήσουμε ότι μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένους κανόνες στους οποίους τα κράτη-μέλη να τηρούν. Υπάρχουν και, άλλες, ε, και άλλα σημεία τα οποία θα ήθελα να αναφέρω προτάσεις δηλαδή που γίνονται για ποινικέ ε, ε, ε, τιμωρίες, για ποινές. Τα ποινικά συστήματα στα κράτη-μέλη είναι τελείως διαφορετικά και το κάθε κράτος μέλος ακολουθεί τη δική του, το δικό του σύστημα. Οπότε δεν μπορούμε να επέμβουμε στο κράτος μέλος και στην ε, ποινική του δικαιοσύνη, αλλά θα πρέπει το σύστημά του ανάλογα με την ε, σοβαρότητα της ποινή, να δίνει, ανάλογα με τη σοβαρότητα του να δίνει και την αντίστοιχη ποινή. Ο ορισμός ε, που υπάρχει λοιπόν για τα δικήματα αυτά και για το, τα παιδιά και για τους ανηλίκους στα κράτη-μέλη είναι τελείως διαφορετικά. Ε, όταν λέμε ανήλικοι μιλούμε για παιδιά κάτω των 18 ετών. Ε, επίσης ένα άλλο καρθόδες ζήτημα είναι το νομικό πρόσωπο. Αν δηλαδή τα νομικά πρόσωπα μπορούν να τιμωρούνται. Και εδώ βλέπουμε πώς ακριβώς, ε, τι, ποιες αντιμετώπισης τη χάνουν οι επιχειρήσεις. οι οποίε θα πρέπει βεβαίω να εφόσον κατηγορούνται ε, και υπάρχουν οι αποδείξει να πληρώνουν όπως ε, με τι ίδιε ποινέ που πληρώνει και ένα φυσικό πρόσωπο. Το θέμα λοιπόν είναι πραγματικά τεράστιο και είναι δύσκολο να, το, να τα πω όλα σε πέντε λεπτά. Απλώς σας ανέφερα τα πιο σημαντικά στοιχεία και ελπίζω η συζήτηση ε, τις επόμενες δύο μέρες να προχωρήσει λίγο παραπάνω. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ε, ευχαριστώ, Πέτρα. Το λόγο έχει η κυρία Γιάννα Κουδάκη που αντιπροσωπεύει την Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φίλων, η οποία εργάζεται πάνω σε μια χνομοδότηση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 Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται να σας αναφέρω όλη την έκθεση γιατί έτσι και αλλιώς έχει δημοσιευθεί. Θα θεωθήξω μόνο κάποιες επιτυχές που είναι πιο επίμαχες. Η κατάχρηση των παιδιών είναι ένα πολύ σκοτεινό γεγονός και είναι πολύ θλιβερό ακόμα περισσότερο όταν παίρνει τη μορφή σεξουαλικής φύσης με εικόνες και χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς η προσωπική διασκέδαση. Η παιδική πορνογραφία έχει αυξηθεί με την ανάπτυξη του ίντερνετ καθώς ε, ε, ενήλικοι και γονεί αλλά και πολιτικοί έχω ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνη για την προστασία όλων των παιδιών. Σε, καθώς ο κόσμος μεταβάλλεται διαρκώς θα πρέπει να μπορέσουμε κι εμείς να εξελιχθούμε και να αντιδράσουμε και να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Εγώ καλωσορίζω τη συνολική πρόταση της ε, Κομισιόν που κατανοεί την, την ανάγκη για μια ολιστική γενική σφαιρική προσέγγιση προστασία, πρόληψη και δίωξη είναι οι λέξεις κλειδιά. Ε, θα ήθελα να αναφέρω μια διατύπωση από την έκθεση και να εστιάσω στους ορισμούς που χρησιμοποιούνται. Τώρα, ο ορισμός της Κομισιόν είναι ότι ένα παιδί είναι κάθε άτομο κάτω από την ηλικία του 18, αλλά κατά την άποψή μου αυτό είναι πολύ ευρύ. Πρέπει να διακρίνουμε ανάμεσα σε ένα παιδί που είναι κάτω από την ηλικία συγκατάθεσης, που, είναι, ποικίλια ποικίλει από χώρα σε χώρα, και τα παιδιά που είναι κάτω των 18 και χρειάζονται προστασία από σεξουαλική εκμετάλλευση ολόκληρη τη γνωμοδότησή μου, όπω και στην πρόταση τη Κομισιόν, χρησιμοποίησα την όρο παιδική πορνογραφία αντί για εικόνες παιδική κατάχρηση παιδιών. γιατί αυτό είναι ένας ευρύτερος όρος που μπορεί να καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα ποινικών πράξεων και όχι απαραίτητο σεξουαλικών. Επιπλέον, όταν εξετάζουμε την ισχύουσα νομοθεσία και ορολογία νομική ορολογία σε συμβάσει που σχετίζονται με αυτήν εδώ τη γνωμοδότηση, είναι πιο συνετό να παραμένουμε στη χρησιμοποιούμενη ορολογία. Βέβαια, αυτό συζητείται για την ώρα. Τώρα, όσον αφορά την πρόληψη, δεν μα έχει διαφύγει το γεγονό ότι ε, μία από τι πιο πολύ συζητημένε πτυχές της τη Κομισιόν είναι για το μπλοκάρισμα και διαγραφή περιεχομένου παιδική πορνογραφία online. Σε αυτό θα πρέπει να είμαστε σαφείς στους στόχου μα. Εγώ ισχυρίζομαι σε συμφωνία με την Επίτροπο Μάλστρομ ότι ο απότερο στόχο είναι να αφαιρεθούν τέτοιου είδου sites μέσω τη ε, διαγραφή του στην πηγή. Αν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν θα πρέπει να είναι δυνατό το μπλοκάρισμα αυτών των ε, site. Αυτό είναι ένα εργαλείο μέσα στο πλωστάσιο που έχουμε. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε όμως ότι τα παιδιά ε, έχουν να αντιμετωπίσουν και τον κίνδυνο ότι κάποιες εικόνες στο ίντερνετ μπορούν να, ε, να τις κατεβάσουν πολλές φορές. Δεν είναι μόνο μία φορά που χρησιμοποιούνται οι εικόνες άπαξε και το περιεχόμενο αυτό δεν είναι απαγορευμένο. Τώρα βέβαια θα πρέπει να στραφούμε και στο θέμα της παιδείας των παιδιών και των γονιών. Η σημασία του κουμπιού πανικού, ε, του ορίου πανικού ε, είναι πολύ μεγάλη. Θα πρέπει να γίνουν, ε, να γίνουν έλεγχοι μέσα στους οποίους θα συμμετέχουν και τα ίδια τα παιδιά. Συχνά ξεχνάμε ότι μεγάλο τμήμα των δραστών μπορεί να είναι και τα ίδια τα, και παιδιά, τα οποία δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο όπως οι ενήλικες Τώρα, σε σχέση με τη δίωξη, πιστεύω ότι η Κομισιόν έχει ξεπεράσει την αρμοδιότητά τη, συμπεριλαμβάνοντα συγκεκριμένου όρου και καταδίκε. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να ορίσουν τι δικέ του ποινικέ κυρώσει. Ωστόσο, μπορεί να αναφέρουμε τι καλύτερε πρακτικέ όταν μιλάμε για καταδίκε. Η δίωξη επίση θα πρέπει να εξεταστεί με τη δυνατότητα αποκατάσταση και με συγκεκριμένα προγράμματα αυτά θα πρέπει να μπορούν να απευθύνονται σε όλους τους ανθρώπους, ε, άσχετα από το αν έχουν αποδεχτεί την ευθύνη τους ή όχι, την ενοχή τους ή όχι. Τώρα, σε σχέση με την οικογένεια του δράστη θα πρέπει επίσης να τη λάβουμε υπόψη, γιατί πολύ συχνά είναι αθώοι άνθρωποι οι οποίοι στιγματίζονται διαβίου λόγω των πράξεων του ενόχου. Ε, εν πάση περιπτώσει η προτεραιότητά μα θα πρέπει να είναι η προστασία των παιδιών και ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη μορφή προστασία. Δεν θα πρέπει να δηλιάσουμε μπροστά σε δύσκολα θέματα όπω το ίντερνετ επί τη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή των ατομικών ελευθεριών και αυτό η οδηγία είναι ένα τομέα όπου μπορεί να υπάρξει δράση εν μέσω μιας ενωμένης προσέγγισης από το σύνολο των κρατών μελών γιατί η οδηγια ειναι ενα τομεα οπου μπορει να υπαρξει δραση εν μεσω μια ενωμενη προσεγγιση απο το συνολο των κρατων μελων γιατι η καταχρηση παιδιων και ε, η παιδική πορνογραφία δεν γνωρίζει σύνορα αυτό και θα πρέπει και εμείς να αντιδράσουμε ενωμένα. Ευχαριστώ τη Μαρίνα και να περάσουμε τώρα στις εργασίες μας αυτές καθε αυτές μετά τις εισαγωγικέ παρουσιάσεις. Να ξεκινήσουμε με την επικεφαλής του γραφείου της Επιτρόπου Μάλστρουμ, η οποία δυστυχώς σήμερα δεν μπόρεσε να παραστεί. Να δώσω λοιπόν το λόγο εξ ονόματο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Μαρία Ασένιους. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much, Madam Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω εδώ σήμερα και θα ήθελα να σας διαβιβάσω τους θερμούς χαιρετισμού της κυρίας Μάλστρομ. Θα ήθελε να βρίσκεται σήμερα εδώ, αλλά δυστυχώς βρίσκεται σε αποστολή εκτός Βερξελών. Η πρόσκλησή σας μου δίνει τη δυνατότητα να σας ε, περιγράψω λίγο το σκεπτικό της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την οδηγία αυτή, για την καταπολέμηση της παιδικής τρομογρα... και της σεξουαλικής κακοποίησης και θα ήθελα να σταθώ σε κάποιες επικρίσεις ε, που γίνονται ενάντια σε κάποιες ε, προτάσεις, κυρίως μια πρόταση που αφορά ε, το ίντερνετ. Δεν χρειάζεται νομίζω να σας πω για ποιο λόγο πρέπει να καταπολεμήσουμε τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την παιδική πορνογραφία. Πρόκειται για σοβαρά παραπτώματα που δημιουργούν μακροπρόθεσμες ε, ζημίες στα θύματα. Είναι αδικήματα τα οποία ε, διαπράττονται κατά των πιο ευάλωτων, των ανθρώπων που είναι πιο ευάλωτοι στην ε, κοινωνία μας, όπως μας υπενθυμίζει η Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αυτών του οποίου τους οποίους έχουμε υποχρέωση να, να στηρίξουμε περισσότερο. Υπάρχουν δεδομένα και ερευνητικά στοιχεία στον τομέα. Δεν θα σταθώ σε αυτά. Θα σας δώσω ένα-δυο στοιχεία για να έχετε μια εικόνα. 10 στα 20 παιδιά μπορεί να βιώσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια μορφή ε, κακοποίησης. Πορνογραφικές εικόνες ή εικόνες ε, παιδικής κατάχρησης όπως αποκαλούνται είναι πάμπολες. Ε, πολλές φορές χρησιμοποιούνται δίκτυα κοινωνικής διοκτήωσης για αποπλάνηση παιδιών και ο σεξουαλικός θερισμός νομίζω είναι γνωστός στη σπάση. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτά τα δικήματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια οδηγία στις αρχές του έτους. Η πρόταση είναι πολύ φιλόδοξη και προσπαθεί να έχει μια συνολική προσέγγιση, να προβλέπει διατάξεις όχι μόνο για τη δίωξη των παραβατών, αλλά ε, και θέματα προστασίας, ε, τα τρία π που ανέφερε η κυρία Γιανακουδάκη μόλις πριν από λίγο. Θα αναφερθώ λοιπόν, λοιπόν σε αυτά, στη δίωξη, στην προστασία και στην πρόληψη. Για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τα θέματα δίωξη, η πρόταση ζητά από τα κράτη-μέλη να προσεγγίσουν την νομοθεσία του και να έχουμε ένα πλήρη κατάλογο ε, περίπου 20 αδικημάτων και να υπάρχουν και αντίστοιχε ποινέ ανάλογα με τη σοβαρότητα του αδικήματο. Ε, καλύπτουν διάφορες μορφές ε, σεξουαλικής κατάχρησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης, κυρίως τις νέες μορφές οι οποίες διαπράττονται πλέον πιο εύκολα λόγω της ανάπτυξης του διαδικτύου. Όπως για παράδειγμα η σεξουαλική παρελέγχληση μέσω διαδικτύου, ε, παιδική πορνογραφία στην οποία έχει πρόσβαση κάποιος χωρίς να πρέπει να κατεβάσει εικόνες που είναι πολύ εύκολο να γίνει σε πολλές χώρες μέλη ε, ορισμένες φορές επίσης έχουμε και κατάχρηση ανηλίκων ζωντανά στο διαδίκτυο μέσω κάμερας. Η αστυνομία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κάνει έρευνες ε, ε, με πολιτικά και να μπορέσει φυσικά να ε, δει αν τηρούνται κάποιες δικλείδες ασφαλείας και κάποιες διαδικασίες. Επίσης, εάν δεν κάνει καταγγελία ένα παιδί ή αν αποσύρει την καταγγελία του θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να συνεχιστεί η ποινική δίωξη και για τα πιο σοβαρά παραπτώματα μπορεί να διωχθούν ε, οι δράστες πολλά χρόνια μετά από τη διάπερξη του για να διασφαλίσουμε ότι αποδίδεται δικαιοσύνη ακόμα και αν τα παιδιά ε, ε, ομολογήσουν τι συνέβη ακόμα και όταν θα είναι πλέον ενήλικες. Επίσης, ε, πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να διωχθούν όταν διαπράττουν αντικείμενα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε το σεξουαλικό τουρισμό. Για το δεύτερο τώρα πει, την προστασία, για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά από την ε, κακοποίηση, θα ενισχύσουμε την πρόσβαση στη νομική συνδρομή και σε ορισμένε περιπτώσεις θα υπάρχει και ένας ειδικό εκπρόσωπος για να βοηθήσει τα θύματα. Θα καθορίζει κανόνες για το πώς θα πρέπει να εκποδεύεται το αστυνομικό και δικαστικό προσωπικό για να κάνει έρευνες με τρόπο που δεν θα τραυματίζει επιπλέον τα παιδιά και η οδηγία αναγνωρίζει ότι πρέπει να γίνουν πάρα πολύ σοβαρές προσπάθειες προκειμένου να διαπιστώσουμε ποια παιδιά έχουν υπάρξει θύματα παιδικής πορνογραφίας και πώς μπορούμε να τα βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν τις τραυματικές εμπειρίες αυτές. Το τρίτο π είναι η πρόληψη. Σαφώς πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε να προλάβουμε όλα αυτά τα δικήματα και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο από τα καθήκοντα που μας αναλογούν το να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά για να μπορέσουν να αναγνωρίζουν πότε μπορεί να υπάρχει κίνδυνος κακοποίηση και κατάχρησής τους ε, ε, είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν μία σειρά από ευρωπαϊκά προγράμματα συμπεριλαμβανομένου και του προγράμματος Δάφνη αλλά ε, η οδηγία προτείνει και άλλα προληπτικά μέτρα μέσα στα πλαίσια φυσικά αυτών που είναι νομικά αποδεκτά μέσω των νομικών μέσων που διαθέτουμε. Καταρχάς, ε, η ειδική μεταχείριση και προγράμματα παρέμβασης έχει διαπιστωθεί ότι έχουν καλά αποτελέσματα και ορισμένες φορές ε, μπορούμε να έχουμε ε, και λύσεις για πολλούς από τους δράστες ή και για άτομα τα οποία δεν έχουν ακόμα διαπράξει κάποιο αδίκημα αλλά μπορεί να υπάρχει κίνδυνος να τη διαπράξουν και χρειάζονται βοήθεια. Δεύτερον, δεν θα ε, για παραβάτε για του οποίου δεν επιτρέπεται κατόπιν καταδίκη να εργάζονται με παιδιά σε ένα κράτο μέλο, δεν θα επιτρέπεται να εργάζονται με παιδιά και στι υπόλοιπε χώρε. Θα υπάρχει μια διαδικασία αμοιβαία αναγνώριση δηλαδή για αυτέ τι εντολέ ε, απαγόρευσης. Και επίσης ε, προσπαθούμε να περιορίσουμε την ε, κυκλοφορία παιδικού περνογραφικού υλικού και εδώ έχουμε την, ε, το άρθρο 21 της οδηγίας το οποίο έχει τραβήξει αρκετή προσοχή ίσως περισσότερο από όσοι χρειάζεται γιατί τα υπόλοιπα 20 άρθρα είναι εξίσου σημαντικά. Να σταθώ όμως λίγο σε αυτό το άρθρο. Η παιδική πορνογραφία και εδώ δεν μιλάμε για εικόνες βιασμένων παιδιών, κακοποιημένων παιδιών ή βρεφών, αλλά γενικότερα παιδικής πορτογραφίας είναι ένα ε, ολαιόν ευξανόμενο πρόγραμμα. Βάσει μιας έκθεσης των ΗΠΑ Κάθε μέρα ανεβαίνουν 200 νέες φωτογραφίες ε, κακοποίησης παιδιών και υπάρχουν εκθέσεις που μας ε, καταδεικνύουν ότι ε, πολλές από αυτές τις εικόνες είναι και πιο βίες και πιο σαφείς ως προς αυτό που δείχνουν. Και οι προσπάθειες που γίνονται και η ευρύτατη διανομή κάνει και πιο επαγγελματική την όλη διαδικασία τα κράτη-μέλη θα υποχρεούνται να αφαιρέσουν το περιεχόμενο παιδικών περιογραφικών εικόνων στην πηγή και να απαγορεύσουν τη ε, λειτουργία ιστότοπων που παρουσιάζουν τέτοιο υλικό το, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν το προτείνει αυτό σαν εναλλακτική λύση, αλλά το προτείνει ως ένα συμπληρωματικό εργαλείο. Και εδώ θα πρέπει να διευκρινίσω το εξή. Δεν υπάρχει θέμα διακοπής της πρόσβασης των χρηστών στο διαδίκτυο. Απλώς δεν θα επιτρέπεται στους χρήστες να κοιτούν τις συγκεκριμένες σελίδες που ε, κυκλοφορούν παιδικό πορνογραφικό υλικό. Το προτιμητέο φυσικά θα ήταν να ε, πατάξουμε το αδίκημα στην πηγή του, αλλά ορισμένες φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί αυτό στην πράξη και σε κάποιες περιπτώσεις είναι και αδύνατο, διότι το παράνομο περιεχόμενο ε, πολλές φορές φιλοξενείται σε ε, ιστότοπους τρίτων χωρών και από μέρα σε μέρα μπορεί να μετακινείται σε διαφορετική χώρα και σε διαφορετική ιστοσελίδα. Ε, φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί με τρίτε χώρε για το θέμα αυτό και η Επίτροπο Μάλστρο το έθεσε και στι Ηνωμένε Πολιτείε και στη Ρωσία προσφάτω. Αλλά παρά τι προσπάθειε όλων όσων ε, ε, συμμετέχουν για να προσπαθήσουν να πατάξουν την παιδική προνογραφία, μόνο με την απαγόρευση, με το blocking αυτών των σελίδων θα μπορέσουμε να περιορίσουμε την κυκλοφορία εικόνων παιδική προνογραφία και έτσι η εμπορία τους θα είναι λιγότερο κερδοφόρα και έτσι ε, θα έχουμε και λιγότερη εκμετάλλευση θυμάτων. Και επίσης με τον ίδιο τρόπο νομίζω θα περιορίσουμε και τον κίνδυνο να το δει κάποιος κατά λάθο ε, όταν ε, σερφάρει στο διαδίκτυο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσβλέπει στη συνεργασία με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών για την προώθηση αυτής της οδηγίας και ελπίζουμε να υιοθετηθεί σύντομα το κείμενο οδηγίας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο Ντανιέλ Φλόρ από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την Προεδρία. Καλώ τους υπόλοιπους προσκεκλημένους να καθίσουν εδώ στο Προεδρείο. Παρακαλώ. την κυρία Φλόρ να πάρει το λόγο. Α, όχι, τον κύριο. Διορθώνει η πρόεδρος. Τον κύριο Φλόρ. Ευχαριστώ κυρία Αντζελίλη. Καταρχήν το Συμβούλιο ευχαριστεί την Επιτροπή σας και σας ιδιαίτερος, κυρία Ισηγήτρια, για την διοργάνωση αυτής της δημόσιας ακρόασης που θεωρούμε ότι είναι πολύ χρήσιμη και σημαντική σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα σε πολιτικό επίπεδο τόσο για τα κρατη όσο και για τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Σε αυτό το στάδιο, όπως γνωρίζετε, δεν μπορώ να σας πω από εξονόματος του Συμβουλίου ποια είναι το, η έκβαση των συζητήσεων μέσα στο Συμβούλιο, γιατί δεν έχουμε ακόμα καταλήξει σε κάποια συγκεκριμένη προσέγγιση σε σχέση με αυτό το εργαλείο. Το θέμα είναι όμως ότι αποτελεί προτεραιότητα για το Συμβούλιο και ιδιαίτερα προτεραιότητα για τη Βελγική Προεδρία. Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η συζήτηση να εξελιχθεί, να προχωρήσει πολύ γρήγορα και να μπορέσουμε επίσης γρήγορα να υποβάλουμε το ζήτημα στο ίδιο το Συμβούλιο και να καταλήξουμε σε μια γενική θέση και να ξεκινήσει έτσι και διάλογο με το Κοινοβούλιο. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, έχουμε σκοπό να πάμε στο Συμβούλιο του Οκτωβρίου ήδη με ένα πρώτο κομμάτι διατάξεων και να επανέλθουμε έπειτα τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο με το σύνολο των ε, διατάξεων ε, και να μπορέσουμε να έχουμε έτσι μια θέση του Συμβουλίου μέχρι το τέλος του έτους για να μπορεί και το Συμβούλιο να μπορεί να μπει σε διάλογο με το Ευρωκοινοβούλιο πριν το τέλος του έτους. Δεν μπορώ να σας πω πιο πολλές λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο. Θα εξαρτηθεί από το ταχύτητα με την οποία θα προχωρήσουν συζητήσεις στο Συμβούλιο. να σας πω λοιπόν καταρχήν ποια είναι τα θέματα τα οποία εξετάζει το Συμβούλιο όσον αφορά την ιδιαιτερότητα αυτού του μέσου και έπειτα να σας υποδείξω κάποια σημεία που αποτελούν πιο δύσκολα σημεία. Καταρχήν, Το Συμβούλιο έχει υπόψη ότι πρόκειται για ένα μέσο αρκετά ε, συγκεκριμένο, δεδομένο το αντικειμένο του. Και υπάρχουν τέσσερα σημεία ε, στα οποία είναι ιδιαίτερα προσεκτικό το Συμβούλιο. Καταρχήν το γεγονός ότι πρόκειται για ένα ε, ε, ποινικό δίκαιο. Και μέσα στα πλαίσια ενός τέτοιου μέσου είναι περιορισμένα τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε υπέρ μιας γενικής προσέγγισης και φυσικά όλες οι διατάξεις ποινικού δικαίου δεν μπορούν να βρουν τη θέση τους σε ένα τέτοιο μέσο ε, ποινικού δικαίου. Είναι πολύ σημαντικό επίση να είμαστε συνεπείς με τα όσα έχουν ήδη γίνει και ιδιαίτερα η διαπόφαση πλαίσιο του 2003 και τη σύμβαση του Συμβουλίου του Ευρώπη ε, του 2007 Λανζαρότε. Δηλαδή είναι βασικό να συνεχίσουμε με βάση τα όσα έχουν ήδη γίνει και να μην υπάρχουν υπαναχωρήσει. Τρίτο σημαντικό στοιχείο και αυτό ήδη το έχουμε τονίσει σήμερα είναι ότι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία είναι η διάσταση των νέων τεχνολογιών και του ρόλου που παίζουν αυτές, ιδιαίτερα το ίντερνετ, στην ανάπτυξη μορφών εγκληματικότητας και μέτρα τα οποία είναι ιδιαίτερα απαραίτητα στον τομέα αυτό για την προστασία των παιδιών. Και τελευταίο στοιχείο είναι αυτό, και αυτό έχει αναφερθεί επίσης, ότι στον τομέα αυτό υπάρχουν διάφορα ε, ε, γεγονότα τα οποία μπορεί να ποινικοποιηθούν. Και ακριβώς αυτό σημαίνει λεπτομερή προσέγγιση όσον αφορά τις ποινές και τα όρια των ποινών που θα προβλεφθούν. Εδώ, λόγω της μεγάλης ποικιλία ε, των ε, αδικημάτων, θα πρέπει να προβλεφθεί αντίστοιχα και μεγάλη ποικιλία ποινών. Αυτά λοιπόν για να σας πω σε ποιους άξονε κινείται η συζήτηση στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Τώρα όσον αφορά τα πιο δύσκολα ε, θέματα, αλλά και πάλι δεν θα σας πω τίποτα καινούριο σε σχέση με αυτά που ήδη υπόθηκαν σήμερα, ένα πρώτο σημείο λοιπόν είναι το θέμα του ορίου μεταξύ του νόμιμου και του παρανόμου, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανάπτυξη της σεξουαλικότητας των εφήβων. Μέχρι πού πρέπει δηλαδή κανείς να ποινικοποιήσει και πού ξεκινά η ελευθερία πειραματισμού των, των εφήβων. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να δούμε ε, πού αρχίζει η ποινικοποίηση. Δεύτερο στοιχείο δύσκολο είναι το θέμα της ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά καταδίκες για αυτού του είδους συμπεριφορές. Εδώ έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο με την ε, διασύνδεση των ε, ποινικών μητρών. Όμως τα συστήματα απαγόρευσης είναι πολύ διαφορετικά στα διάφορα κράτη-μέλη και δεν είναι πάντοτε συμβατά. Γι' αυτό και είναι δύσκολο να ε, ισχύσει ένα παρόμοιο σύστημα σε όλα τα κράτη-μέλη, γιατί ανάλογα με τα μέτρα που προβλέπονται, είτε αυτά είναι αστικού δικαίου, είτε είναι διοικητικού, είτε είναι ποινικού, οι ποινέ μάλλον που προτείνονται είναι πολύ διαφορετικές και έτσι η αναζήτηση κοινών λύσεων καθίσταται πολύ δύσκολη. Το σημαντικό σημείο και δύσκολο σημείο είναι η δικαιοδοσία υπάρχει βούληση να καλυφθεί ο σεξουαλικός τουρισμός και άρα ανάγκη αρμοδιότητα αρμοδιότητας αρκετά ευρεία, όμως ταυτόχρονα αυτές οι εξοεδαφικές αρμοδιότητες θα πρέπει να μπορούν να εναρμονίζονται με τις τεράστιες διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα νομικά συστήματα των κρατών μελών. Δυσκολία δηλαδή εξέβρεση ισορροπία ανάμεσα στη βούληση να προχωρήσουμε με κατάλληλο τρόπο στι εξωτερικέ υποθέσει όπω αυτέ του σεξουαλικού τουρισμού και ανάγκη να εντασσόμαστε πάντα μέσα στο πλαίσιο των νομικών συστημάτων των κρατών μελών. Ταυτόχρονα το θέμα, το θέμα του μπλοκαρίσματος των site. Υπάρχουν διαφορές στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν υπόψη τα στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμα και έπειτα υπάρχουν και τεχνικές πτυχές. Μπορεί να πάρουμε μέτρα τα οποία είναι πολύ ωραία και καλά στο χαρτί, αλλά ποιες είναι οι δυνατότητες σε τεχνικό επίπεδο. Σημαντικά μέτρα λοιπόν, τα οποία όμως δημιουργούν ε, ερωτήματα σε τεχνικό και νομικό επίπεδο. Η Προεδρία περιμένει λοιπόν να προχωρήσει η συζήτηση στο πλαίσιο του Συμβουλίου και θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι είμαστε αποφασισμένοι να φέρουμε σε αίσιο πέρας τη συζήτηση σε αυτό το χρόνο και μάλιστα μέσα στο, πριν το τέλος μάλλον της Προεδρίας μας. Δηλαδή πριν το τέλος του χρόνου. Ευχαριστώ. Merci, Σας ευχαριστώ κύριε Φλόρα και ευχαριστώ για τη δέσμευση που αναλάβατε εξ ονόματος Συμβουλίου. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Σάρμα, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας διατρέχω τον κίνδυνο να επαναλάβω αυτά που είπαν οι προηγούμενοι, οπότε δεν θα αναφερθώ καθόλου σε αυτά που ακούστηκαν ήδη. Στον, ε, στην Ευρώπη του 21ου αιώνα είναι κρίμα που τα παιδιά μας δεν είναι ασφαλή όπου και να βρίσκονται στον πλανήτη αυτό. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Επιτροπή και η Κοινωνική Επιτροπή, τη οποία είμαι εγώ ε, συγκήτρια για το έγγραφο αυτό, προφανώ καταδικάζει οποιαδήποτε σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών και χρησιμοποιούμε την ε, κοινωνία των πολιτών και εμπειρογνώμονες από αυτήν ώστε να ε, συντάξουμε μία γνωμοδότηση που θα διακατοπτρίζει τι απόψει τη ε, κοινωνία των πολιτών. Η σοβαρότητα τη ποινή, η οικογένεια, το σπίτι, η ευαισθησία των παιδιών δεν θα πρέπει να υπονομεύονται ποτέ. Και γι' αυτό θα πρέπει να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη που δεν έχουν επικυρώσει ακόμη την Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών έναντι της σεξουαλικής κακοποίηση και εκμετάλλευση και το ε, ε, πρωτόκολλο από την CRC ε, του, των Ηνωμένων Εθνών να το υπογράψουν. Αυτό δεν θα πρέπει να το ξαναζητήσουμε έτσι ώστε να μπορέσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπογράψει αυτά τα έγγραφα ε, και τις συμβάσεις όπως έκανα με την συνθήκη της Λισαβόνα. Έχουμε κάνει πολλά σχόλια για συγκεκριμένα άρθρα στα πλαίσια της οδηγίας που θεωρούμε ότι θα πρέπει να τύχουν μεγαλύτερη προσοχή, αλλά θα ήθελα να σχολιάσω κι εγώ κάποια. Καταρχήν, η, η πρόληψη είναι εκ των όνων κάνευ. Ε, θα πρέπει να το δούμε από κοινού με την ομοθεσία. Αυτό ήταν ένα από του βασικού στόχου τη οδηγία. Οπότε πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα στον τομέα αυτό με την βοήθεια και της κοινωνίας των πολιτών και των μηχανισμών που διαθέτει. Χρειαζόμαστε μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών που θα απαντούν σε κάποια από αυτά τα ε, εγκλήματα και νομοθετικά και μη νομοθετικούς ε, μηχανισμούς ώστε να έχουμε μεθοδολογικά εργαλεία και κατάρτιση. Αυτό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τους οργανώσεις της, τις, ε, τους κοινωνικούς εταίρους, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις ώστε να, να υποστηριχθεί η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση σε τοπικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Επιτροπή καλεί και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και την Κομισιόν που έχουν ε, την ε, δεσπόζουσα θέση να ε, επιβάλλουν τους κανόνες αυτούς στα κράτη-μέλη τους και κυρίως τους, τους εταίρους μας που είναι ιδιαίτερα συντηγμένοι, Αυστραλία, Ρωσία, Κίνα, Ιαπωνία, Αμερική, για την αφαίρεση, διαγραφή τέτοιων ιστοσελίδων που έχουν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το σπίτι μας ο καθένας, γιατί η Ευρώπη έχει υψηλό επίπεδο τέτοιων ιστοσελίδων με τέτοιο υλικό. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να υπάρχουν. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γιατί δεν κατεβαίνουν από το ίντερνετ αυτέ τι σελίδε δυνάμει και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και η ΟΚΕ, όπως και οι υπόλοιποι, θέλουμε να αποφερεθούν αυτές οι σελίδες ή τον μπλοκάρισμα των σελίδων αυτών θα πρέπει να γίνεται μόνο αν δεν μπορούν να διαγραφούν. Επίση θα πρέπει να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για την ε, ελάχιστη ηλικία ε, για, το, για τη συγκατάθεση, για να δίνουν τα παιδιά τη συγκατάθεσή τους σε ε, σχέσει ε, σχέσεις ε, σε όλη την Ευρώπη. Είναι ένα θέμα πολύ δύσκολο και πρέπει να υπάρξει ευρεία διαβούλευση για αυτό. η και επίση αναγνωρίζει ότι η Κομισιόν θα πρέπει να δει λίγο του ορισμού που χρησιμοποιεί και εδώ θα ήθελα να δώσω κάποια παραδείγματα. Για... Βέβαια, ακούστηκαν ήδη αρκετά. Ο όρο παιδική πορνογραφία παιδική πορνογραφία θα πρέπει να αντικατασταθεί από, την, ε, από το υλικό ή φωτογραφίες ε, ε, παιδικής εκμετάλλευσης. Η πορνογραφία συνδέεται με το ερωτισμό. Εμείς δεν μιλούμε για ερωτισμό εδώ. Επίσης, σεξουαλικός τουρισμός. Ο σεξουαλικός τουρισμός ο τουρισμός μάλλον συνδέεται με, με διακοπές, με απόλαυση, με ξεκούραση. Θα πρέπει να μιλήσουμε για Αυτού που διαπράττουν σεξουαλικά εγκλήματα και που ταξιδεύουν από χώρα σε χώρα. Πρέπει λοιπόν να δούμε και την επίδραση των παραδόσεων σε αυτό το τομέα. Και εδώ ας πούμε μπορεί να μιλούμε για αφροτηριασμό των γενικών γεννητικών οργάνων που δεν καλύπτονται από την οδηγία. Επίσης πρέπει να δούμε μια, έναν ε, ενιαίο χρονικό ορισμό, περιορισμό. Η ΟΚΕ ζητά το, οι περιορισμοί να ξεκινούν όταν το θύμα φτάνει στην, α, στην ηλικία των 18 και όχι από όταν έγινε η ε, κακοποίηση. Ε, υπάρχουν πάρα πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες λειτουργούν και δουλεύουν για το θέμα αυτό. Υπάρχουν λοιπόν πολλά στοιχεία και, οι, και πολλές μη κυβερνητικέ προσπαθούν να προστατεύσουν τα παιδιά σε όλο τον κόσμο και το και ο ΙΕ και ε, το Συμβουλίο της Ευρώπης προσπαθούν να βρουν τέτοιε τέτοιες διόδους και εργαλεία για να προστατευτούν τα παιδιά σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα ακόμα, δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε άλλες δικαιολογίε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Κοινοβούλιο που μας συμπεριέλαβε στη σημερινή συζήτηση γιατί η φωνή της κοινωνίας των πολιτών είναι σημαντική. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο στην κυρία Μαρία Αμόρ Εστεμπάνεθ, η οποία εκπροσωπεί ε, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου καταρχάς να ευχαριστήσω την Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων που ε, κάλεσε τον Οργανισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εδώ να συμμετάσχει σε αυτή τη συνεδρίαση για να συζητήσουμε την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών και της παιδικής πολλογραφίας. Το περιεχόμενο είναι ευπρόσδεκτο από τον οργανισμό μα, Επί τη βάση σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης και παιδική προνογραφία είναι ε, σαφή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρόκειται για ένα βήμα περαιτέρω για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα από του τομεί, ο οποίος ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον οργανισμένο ε, καθώ τα δικαιώματα των παιδιών αποτελούν ε, μία από τι βασικέ θεματικέ ονότητε του οργανισμού στο πολιτέ τη πρόγραμμα υπηρεσία ε, προσπαθεί να εργαστεί σε θέματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Βασιζόμαστε σε δύο άρθρα της συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 67 που καθορίζει την υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ε, διασφαλίζει ψηλό επίπεδο ασφάλειας για την καταπολέμηση αδικημάτων και το άρθρο 83 μέσω του, του οποίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να καθορίσουν ελάχιστους ε, κανόνες για ποινικά δικήματα και κυρώσεις για πολύ σοβαρά δικήματα τα οποία έχουν διαμεθοριακή διάσταση. Η πρόταση επίσης αναφέρεται και στη σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών ως κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Ε, πρόκειται για μια πολύ σοβαρή μορφή εγκλήματος και φυσικά τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε ειδική φροντίδα. Και όλα αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όπως επίσης ε, η η προστασία των παιδιών που αναγνωρίζεται στο άρθρο 24 της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, βάσει του οποίου τα παιδιά θα πρέπει να προστατεύονται, διότι αυτό είναι απαραίτητο για την ευημερία τους και ε, οι κυρώσει είτε λαμβάνονται από ε, οι δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ε, θα πρέπει να έχουν ως πρώτο μέλημά τους την φροντίδα των παιδιών. Η νέα συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πλέον αναφέρει ρητά την υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προστατεύει τα παιδιά και φυσικά στην απόφαση του δικαστηρίου της 27ης Ιουνίου του 2006 στην υπόθεση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά του Συμβουλίου ε, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ε, Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας ε, η Σύμβαση των Δικαιωμάτων των Παιδιών πρόκειται για ένα από τα μέσα προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων το οποίο λαμβάνει υπόψη την εφαρμογή των βασικών αρχών του κοινοτικού δικαίου. Όλα τα κράτη-μέλη ε, επίσης ε, συμμετέχουν στη διάσκεψη για τα δικαιώματα των παιδιών για την παιδική πορνογραφία και την παιδική πορνεία, παρά το γεγονος οτι ότι κάποια κράτη-μέλη δεν το έχουν ακόμα κυρώσει και περιμένουμε και ανάλογη απόφαση του δικαστηρίου για το πρωτόκολλο αυτό. Επίσης δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Συμβουλίου για την σεξουαλική προστασία και τη σεξουαλική κακοποίηση έχει υπογραφεί προσφάτως από την πλειονότητα των κρατών μελών και η κύρωση προχωρά με πολύ καλό ρυθμό. Η ενεργή συμμετοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών στον τομέα αυτό θεωρείται πλέον απαραίτητη συνθήκη. Αυτό που είναι σημαντικό επίση είναι να έχουμε συνέπεια με πολιτικέ και στόχους Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά το δικαίωμα να σεβαστούμε την ιδιωτική και δημόσια ζωή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όπω βάσει και του άρθρου 8 το χάρτα των θεμολογικών δικαιωμάτων και των άρθρων 7 και 8 Επίσης αναφερόμαστε και στην ελευθερία της έκφρασης τη Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το άρθρο 11 τη χάρτα χρειαζόμαστε να έχουμε μία ε, δράση εξισορρόπησης για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι έχουμε προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επίσης αναφερόμαστε στην αξιολόγηση αντικτύπου που έγινε από την προηγούμενη απόφαση για φιλικό διακανονισμό της 29 η Μαρτίου του 2009 με τον ίδιο τότλο και θεωρείται ότι ισχύει η μουτά τη μουτάντη και για την παρούσα πρόταση. Επειδή όμω η πρόταση αυτή ε, περιλαμβάνει πολλά σημαντικά νέα στοιχεία, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι σε πολλά νέα κράτη-μέλη έχουμε κυρώσεις και υποχρέωση από πλευράς κρατών μελών να λαμβάνονται μέτρα για να αφαιρούνται από το διαδίκτυο εικόνες που παρουσιάζουν παιδική πορνογραφία ε, και η σημασία αυτών των μέτρων απαιτεί να γίνει μια πολύ ε, καλή αξιολόγηση αντικτύπου. Οι νέες τεχνολογίες και κυρίως το διαδίκτυο θα πρέπει ε, να σέβονται τις διατάξεις για την ελευθερία του λόγου και φυσικά θα υπάρχει η ανάλογη προστασία. Θα πρέπει, βάσει του κράτου δικαίου, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι να καθορίσουν τι είναι παραβίαση των δικαιωμάτων των υπολείπων και τα μέλη του δικαστικού και αστυνομικού κλάδου που είναι υπεύθυνα για την ε, προστασία κατά των αδικημάτων ε, να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχουν παραβίαση κατά τη ιδιωτική ε, ζωή όταν έχουμε περιεχόμενο το οποίο είναι κατά τη ζωή των άλλων. Η απόφαση του Δικαστηρίου για την ερμηνεία των άρθρων 10 και 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης ε, καθορίζει σαφώς τι θα πρέπει να θεωρείται περιεχόμενο το οποίο ε, παραβιάζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων. Οι δικαιοργανώσεις ε, οι οποίες θα πρέπει να δρούν ως επόπτες για να διασφαλίσουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρίνεται καταλήλως και δεν γίνεται κατάχρηση είναι πάρα πολύ σημαντικές και θα πρέπει να παραμείνουν όσοι έχει στο μέλλον. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το δικαίωμα ελευθερία έκφραση δεν παραβιάζεται μέσω παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων όσων ερευνούνται για παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών, ε, συμπεριλαμβανομένη και τη χρήση του δικτύου και των νέων τεχνολογιών. Η πρόταση επίσης αναφέρει ότι ε, σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει ε, εσκεμμένη συμπεριφορά του δράστη και θα πρέπει να ε, καθορίσουμε τι σχέση υπάρχει μεταξύ της χρήσης του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών εν γέννη και το θέμα είναι ότι η χρήση του διαδικτύου ορισμένες φορές δίνει τη δυνατότητα σε κάποιους ανθρώπους να καταχραστούν άλλους που δεν έχουν τις τεχνικές γνώσεις να γνωρίζουν τι γίνεται στο διαδίκτυο. Επίσης υπάρχουν απαιτήσει ε, να υπάρχει πρόσβαση εν γνώση ε, του οποιοδήποτε. Το άρθρο 10 της πρότασης ασχολείται με τις καταδίκες και αυτό προσπαθεί να προλάβει την επανάληψη των ίδιων ε, αδικημάτων και αυτό προκύπτει από το άρθρο 7.1 και 7.2 της απόσαφασης του 2009 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το περιεχόμενο και την ανταλλογή πληροφοριών τα οποία προκύπτουν από ποινικά μητρώα μεταξύ κρατών μελών. Μπορούμε να περιορίσουμε τον ε, τύπο των προσωπικών δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και φυσικά αυτό μπορεί να συνεισφέρει για να έχουμε περισσότερες δικλείδες ασφαλείας για την ιδιωτική ζωή των ανθρώπων που ε, συμμετέχουν σε τέτοια δικήματα. Επίσης, όσοι τα δικάζονται για συγκεκριμένα δικήματα πρέπει να προστατεύονται ε, βάσει του άρθρου 20 της πρότασης. Όσον αφορά τώρα τη συνένεση, τη συγκατάθεση κάποιων ε, για συγκεκριμένα προγράμματα ή μέτρα, η παράγραφος 3 του άρθρου 20 καθορίζει υποχρέωση των κρατών μελών να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι όσοι καταδικάστηκαν από συγκεκριμένα, για συγκεκριμένα δικήματα και μετά ε, στην παράγραφο D συγκατατίθενται γνωρίζοντας ε, συγκεκριμένα γεγονότα μπορεί να αρνηθούν και να μην γνωρίζουν τις ε, δυνητικές συνέπειες μιας άρνησης. Η συμμετοχή των κρατών μελών θα πρέπει να προβλεφθεί για την ανταλλαγή πληροφοριών βάσει ε, του δράστη, ώστε να μπορέσει ε, όποιος λαμβάνει αποφάσεις να λαμβάνει ενημερωμένες αποφάσεις. Η προστασία των θυμάτων θα πρέπει να είναι η βασική μας μέρημνα και θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί που θα μας επιτρέψουν να λάβουμε υπόψη μας αυτό το γεγονός. Και όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται βάσει της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσώπων. Όσον αφορά τώρα τις ποινικέ διαδικασίες και έρευνα, ε, το άρθρο 19 παράγραφος 1 προβλέπει τον ορισμό ενός ειδικού αντιπροσώπου για το παιδί θύμα. Αυτό δεν θα πρέπει να ισχύει μόνο όταν πρόκειται για συνόδευτο ανήλικο από, τους, ε, από τα μέλη της οικογένειάς τους, αλλά και για παιδιά τα οποία έχουν χωριστεί από τους γονείς τους ή τους κηδεμόνες τους. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 19 δεν είναι σαφές αν η διατύπωση μας ε, αναφέρεται στην ανάγκη να υπάρχει συνέντευξη με το παιδί ή αναφέρεται στο γεγονός ότι η συνέντευξη θα πρέπει να γίνεται σε χώρο κατάλληλα προσαρμοσμένο για τα παιδιά. Τέλος, το άρθρο 21 που αφορά το μπλοκάρισμα της πρόσβασης σε ιστοσελίδες που περιέχουν παιδική πορνογραφία δεν κάνει διάκριση μεταξύ διαδικτύου και άλλων ε, τρόπων ε, μετάδοσης παιδικής πορνογραφίας και πρέπει να μην γίνεται διάκριση μεταξύ υλικού που παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων. Οποιαδήποτε μπλοκάρισμα πρόσβασης ε, θα πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει το δικαίωμα των χρηστών ε, να χρησιμοποιούν ελεύθερα ε, το διαδίκτυο και να εκφράζονται ελεύθερα. Θα πρέπει να υπάρχει πιο ακριβή διατύπωση, για παράδειγμα αντικαθιστώντας την ανάγκη να διασφαλίσουμε ότι το μπλοκάρισμα περιορίζεται στα απαραίτητα ε, με το, την ανάγκη να διασφαλίσουμε ότι το μπλοκάρισμα περιορίζεται ε, σε υλικό παιδικής πορνογραφίας, διασφαλίζοντας ότι μόνο το υλικό παιδικής πορνογραφίας θα διακόπτεται, θα απαγορεύεται στο διαδίκτυο. Ε, έτσι ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα κάποιος να ε, προσβάλλει το γεγονός ότι μπλοκαρίστηκε μία ε, σελίδα στο διαδίκτυο. Διότι έτσι όπως αναφέρεται στην πρόταση δεν είναι σαφές και θα μπορούσαν να υπάρξουν παρερμηνίες. Θα ήθελα ολοκληρώνοντας να πω ότι η πρόταση είναι πολύ σημαντικό μέσο όχι μόνο για την ενίσχυση του ποινικού δικαίου αλλά και για την προστασία των παιδιών. Ο οργανισμός μας προσβλέπει λοιπόν στην έγκριση της σχετικής οδηγίας και πιστεύουμε ότι θα πρέπει κατά περιόδου περιόδου να παρακολουθούμε και να αξιολογούμε την εφαρμογή τη οδηγία, ώστε να μην υπάρχουν αρνητικέ συνέπειες για τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στα πλαίσια τη εντολή τη, ε, ε, η υπηρεσία θα παρακολουθεί στην εφαρμογή τη οδηγία επιτόπου σε συνεργασία με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά ε, θεσμικά όργανα και οργανισμούς και φυσικά θα παρέχουμε κάθε βοήθεια που είναι απαραίτητα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. E Σας ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους ομιλητές να στείλουν στη γραμματεία της Επιτροπής τις παρεμβάσεις τους γραπτός έτσι ώστε να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όταν θα χρειαστεί να συντάξουμε την ε, πρόταση έκθεσης. Γιατί έχουμε και μάλιστα λιγοστό χρόνο και κάθε ένας από τους ομιλητές χρειάστηκε να είναι πιο συνοπτικός, να μην τα πει όλα αναλυτικά όσα ήθελε να πει. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ζητήσω να γίνει αυτό για τις τεχνικές παρεμβάσεις, όπως έκανε τώρα η υπηρεσία για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Γιατί μας είπατε πολύ συγκεκριμένα πράγματα και αυτό το θέλαμε και γραπτός, για να μπορέσουμε να δουλέψουμε και καλύτερα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπουταρέλη, που αντιπροσωπεύει τον οργανισμό προστασίας δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αγαπητή εισηγήτρια, αγαπητοί κύριοι βουλευτές. Από το σημειώσουμε και από το έγγραφο που έστειλα ήδη στη γραμματεία ΛΥΜΠΕ θα μπορείτε να δείτε πόσο πολύ συμβάλλει ο επόπτης, ο Ευρωπαίος επόπτης ε, ε, των στοιχείων στην καλύτερη προστασία των στοιχείων των παιδιών μέσα στην ε, αυτή κοινωνία της πληροφορίας, όχι μόνο σε σχέση με την παιδική πορνογραφία, αλλά επίσης όσον αφορά τα κοινωνικά δίκτυα, για παράδειγμα η συγκατάθεση παιδιών και γονιών αλλά και η παρενόχληση στο δίκτυο. Να σας πω ότι εκτιμούμε αυτή την πρωτοβουλία που στόχο έχει την ενίσχυση των προληπτικών και των κατασταλτικών μέτρων κατά της σεξουαλικής κατάχρησης και εκμετάλλευσης. Δυστυχώς αυτό το φαινόμενο δεν φαίνεται να μειώνεται. Κατευθύνεται κατά παιδιών που είναι όλα ένα πιο ευάλωτα online και τα οποία έχουν ένα δικαίωμα σε ειδική προστασία και φροντίδα όπως αυτό είναι απαραίτητο για την ε, ευημερία τους. Συνέβαλα ιδιαίτερα στην σύνταξη ειδική νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο. Γι' αυτό και θα ήταν ευπρόσδεκτη σήμερα η δημιουργία ελάχιστων κανόνων σε σχέση με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των ε, κυρώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την εισαγωγή νέων ερευνητικών εργαλείων, καθώς και οποιοδήποτε άλλο άλλη στεναρή κοινωνική απάντηση για να αντιμετωπιστούν νέες μορφές κατάχρησης και εκμετάλλευσης. Επίσης λοιπόν για τον Ευρωπαίο επόπτη το, τα, τα συμφέρον του παιδιού θα είναι το πρωταρχικό του μέλημα. Και γι' αυτό τώρα δεν μιλώ ούτε για την πιθανή ποινικοποίηση νέων ή σχετικά ή μάλλον σοβαρών μορφών κατάχρησης που τιμωρούνται ελαφρά ή σχετικά με την αναγνώριση ειδικών ερευνητικών τεχνικών. Επίσης, η σημερινή μα συμβολή δεν εστιάζει την προσοχή στην εγκυρότητα των αποδείξεων, στην απαγόρευση ορισμένων δραστηριοτήτων, την ανταλλαγή πληροφοριών, στην αδιασφαλιστή εφαρμογή through ε, σε ολόκληρη την Ένωση και νέους κανόνες σε σχέση με τη δικαιοδοσία, τα νομική αντιμετώπιση, τη βοήθεια προς τα θύματα. Εμείς ασχολούμαστε με τις διατάξεις πιο άμεσα που αφορούν μάλλον πιο άμεσα την προστασία προσωπικών δεδομένων και όλος ιδιαίτερος το μπλοκάρισμα πρόσβασης σε ορισμένα sites από τους ε, χρήστες. Υπάρχουν διάφορα δικαιώματα που παραβιάζονται μέσω της σεξουαλικής ε, κατάχρησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών εκτός από την παραβίαση θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων ε, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε νέα νομοθετικά μέτρα θα είναι απόλυτα συμβατά με καμιά νέα φαιά περιοχή και σε απόλυτα συμβατά με τα υπόλοιπα θεμελιώδη δικαιώματα. Εμείς ε, ασχολούμαστε με όλες τις πρωτοβουλίες που έχουν αντίκτυπο στο ρόλο του ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου της επιβολής του νόμου σε σχέση με τον περιορισμό πρόσβασης σε site ε, παιδικής πορνογραφίας δεν αμφισβητούμε την ανάγκη να δημιουργηθεί καλύτερο πλαίσιο που προβλέπει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μειωθεί κυκλοφορία του υλικού αυτού. Ωστόσο, ορισμένα από τα μέτρα που προβλέπονται σε αυτή την πρόταση, όπως η αφαίρεση, η διαγραφή μάλλον ή το μπλοκάρισμα διαφόρων site, καθώς και η δημιουργία ε, ειδικών ε, γραμμών, έχουν αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων των διαφόρων ε, εμπλεκόμενων ατόμων. Ε, ένας μηχανισμός που μπορεί να μπλοκάρει τέτοια, ε, την πρόσβαση σε τέτοια site ή μπορεί να είναι ε, εκούσιες δράσεις για το μπλοκάρισμα ενό site επί τη βάση ενός κώδικα δεοντολογίας. Εμείς θα μπορούσαμε να στηρίξουμε ενέργειες στις οποίες προφέρνει η αστυνομία ή οι δικαστικές αρχές μέσα σε ένα πολύ καλά καθορισμένο νομικό πλαίσιο με πλήρη σεβασμό του νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς και των παραδόσεων που είναι κοινέ στα κράτη-μέλη ιδιαίτερα όσον αφορά την ελευθερία επικοινωνίας και σε σχέση με την στις δικαιοδοσίες που παρέχονται από τα συντάγματα. Έχουμε κάποιες αμφιβολίες όσον αφορά την νομική βεβαιότητα μπλοκαρίσματος που μπορεί να το κάνει κάποιος ιδιωτικός φορέας. Το μπλοκάρισμα μπορεί να σημαίνει διάφορες δραστηριότητε υποπτήρες συμπεριλαμβανομένου του σκάνινγκ του ίντερνετ, εντοπισμό ε, παράνομων ύποπτων ε, ιστοτόπων ή μπλοκάρισμα χρήσης πρόσβασης στους τελικούς χρήστες αλλά και παρακολούθηση των τελικών χρηστών που προσπαθούν να αξιολογήσουν και να κατεβάσουν τέτοιο είδους υλικό. Η πρόταση της Κομισιόν δεν αναθέτει τα ISP με αρμοδιότητες παρακολούθησης παρά μόνο με αρμοδιότητες μπλοκαρίσματος. Ωστόσο, το θέμα είναι πώς θα προβούν σε κάτι τέτοιο χωρίς να παρακολουθούν τους χρήστες. Και αυτό είναι κάτι νέο σε σχέση με την σύμβαση του Συμβουλίου 201 κάθετος 2007. Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν είναι διαφορετικά. Ας πούμε, ε, Έχουμε μπλοκάρισμα DNS, ε, ε, μπλοκάρισμα διευθύνσεων ή και εποπτεία ε, διαφόρων πακέτων. Σημαίνει αυτό διάφορους βαθμούς παρέμβασης και προκαλούν, προκαλεί ερωτήματα όσον αφορά τον ρόλο των ε, προμηθευτών υπηρεσιών στο ίντερνετ σε σχέση με την επεξεργασία του περιεχομένου και της πληροφορίας. Τα προσωπικά δεδομένα διαφόρων ανθρώπων θα εξεταστούν, είτε είναι πληροφορίες για θύματα, είτε είναι για μάρτυρες, είτε για χρήστες ή για τους προμηθευτές περιεχομένου. Δύο βασικές λοιπόν ανησυχίες έχουμε. Η παρακολούθηση του δικτύου και το μπλοκάρισμα site θα αποτελούσε ένα έργο το οποίο δεν σχετίζεται με τον εμπορικό ε, στόχο των προμηθευτών ε, των υπηρεσιών στο ίντερνετ. Δεύτερον, θα ήταν πολύ σημαντικό να υπαλληθεύσουμε καλύτερα αν το μπλοκάρισμα των site θα είναι στο μέλλον ένα αποτελεσματικό μέτρο ή τελικά ένα άχρηστο μέτρο που εύκολα μπορεί να παρακαμφθεί. Ποια είναι τα κριτήρια για το μπλοκάρισμα, ένα κώδικα διοντολογία ή κάποιε εκούσιε κατευθύνσει γραμμέ. Αυτά δεν θα έδιναν επαρκή νομική βεβαιότητα. Έπειτα, οι κίνδυνοι που συνδέονται με την πιθανή μαύρη λίστα ατόμων και τις δυνατότητες τους αποκατάστασης ενώπιον μιας ανεξάρτητης αρχή είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Άρα λοιπόν, αν λάβουμε υπόψη αυτή την παρέμβαση, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι χρειάζονται περισσότερες διασφαλίσεις και γιατί η παρακολούθηση και το μπλοκάρισμα θα πρέπει να γίνονται με αυστηρό δικαστικό έλεγχο και ο μηχανισμός αυτός θα συνοδεύεται από διάφορα μέτρα ασφαλείας. Άρα η αναφορά στο άρθρο 21 στις κατάλληλες ε, ασφαλιστικές ε, δικλείδες ε, είναι αξιέπαινη και είναι μια πρώτη βάση για περαιτέρω ανάλυση. Δεν λέμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει έλεγχο ή μπλοκάρισμα, απλώς ότι θα πρέπει να πλαισιώνεται πολύ σοβαρά. Εκτιμούμε το γεγονό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσφατα σε άλλο πλαίσιο υιοθέτησε όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, ε, υιοθέτησε μια γραπτή δήλωση που στηρίζει την ίδια άποψη. Κάποια τελικά σχόλια όσον αφορά τη δημιουργία ενός, ενός δικτύου ε, γραμμών τηλεφωνικών γραμμών βοήθειας. Αυτό δεν αναπτύσσεται στην ίδια την πρόταση, αλλά αναφέρεται σε ένα προηγούμενο έγγραφο, δηλαδή το πρόγραμμα για ασφαλέστερο ίντερνετ, το οποίο έχουμε ήδη σχολιάσει. Εμείς ε, σχολιάσαμε τις, τους όρους υπό τους οποίους θα μπορούσαν να συγκεντρώνονται αυτές οι πληροφορίες και να ανταλλάσσονται. Από την άποψή μας υπάρχει ανάγκη για συγκεκριμένη περιγραφή του τι θα πρέπει να θεωρηθεί ως παράνομο ή βλαβερό περιεχόμενο Ποιος μπορεί να το συλλέξει, να συλλέξει και να κρατήσει αυτές τις πληροφορίες και ε, σύμφωνα με ποιες συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλείδες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό αν σκεφτεί κανείς ε, τις ε, συνέπειες των αναφορών αυτών. Ιδιαίτερα όσον αφορά τα παιδιά, τα προσωπικά στοιχεία οποιοδήποτε ατόμο που σχετίζεται με πληροφορίες που κυκλοφορούν στο ίντερνετ θα μπορούσε να διακυβευτεί συμπεριλαμβανομένων για παράδειγμα πληροφοριών για ένα άτομο το οποίο είναι ύποπτο για κακή συμπεριφορά. Είτε είναι χρήστη του ίντερνετ είτε είναι προμηθευτή της ε, περιεχομένου ή το ίδιο το θύμα της κατάχρησης. Τα δικαιώματα λοιπόν όλων αυτών των ανθρώπων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα για την προστασία των στοιχείων. Πιθανότατα δε, τέτοιου είδους πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της, δίωξη της και της εισαγγελική έρευνας. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν κατάλληλες ασφαλιστικές δικλειδές ώστε να εγγυηθούνται ότι αυτές οι πληροφορίες που θεωρούνται ψηφιακοί και αποδείξεις έχουν συλλεγεί με το σωστό τρόπο και άρα είναι αποδεκτές και στέκουν σε ένα δικαστήριο. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα λοιπόν διαφάνεια και ανεξάρτητης αποκατάσταση. Υπάρχει ανάγκη λοιπόν εξασφάλιση τη νομική βεβαιότητα για όλα τα μέρη και για τους προμηθευτές του ίντερνετ αλλά και τους, για τους χρήστες με σαφές όπως είπαμε νομικό πλαίσιο και υπάρχει υποχρέωση για τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν μια πραγματικά εναρμονισμένη ε, διαδικασία με όλες τις λεπτομέρειες όταν αφορά, όσον αφορά το παράνομο περιεχόμενο και την εποπτεία ανεξαρτήτων δημοσίων αρχών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Έχουμε τώρα δύο παρεμβάσεις από πλευράς ε, δύο συναδέλφων. Επίσης, σας ζητώ να σεβαστείτε λίγο το χρονοδιάγραμμα γιατί έχουμε μια μικρή καθυστέρηση. Η κυρία Ινετφέλτ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομη. Uh, Χαίρομαι για τις δράσεις που λαμβάνονται κατά της ε, σεξουαλικής εκμετάλλευσης και όλων αυτών των των πράξεων που συζητάμε σήμερα. Αλλά αν κάνουμε κάτι τέτοιο θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι είναι αποτελεσματικά αυτά που κάνουμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Στη διάρκεια της συζήτησης ε, και των παρουσιάσεων που ακούσαμε σήμερα το απόγευμα θα ήθελα να πω ε, και να χρησιμοποιήσω μια βρετανική έκφραση που μου αρέσει πάρα πολύ. Υπάρχει ένας γορίλας 300 ε, κιλών εδώ στην αίθουσα. Αναφερόμαστε σε όλους τους ματάκιδες εντός εισαγωγικών που πριν κρυβόντουσαν στους τάβνους και τώρα είναι στο διαδίκτυο ξεχνάμε ότι το 80% των περιπτώσεων σεξουαλικής εκμετάλλευσης δεν γίνονται από εγκληματίες αλλά από ανθρώπους στο κοντινό οικογενειακό του περιβάλλον, στο σχολείο, στο σπίτι, στα αθλητικά κέντρα και στις εκκλησίες. Πλέον είναι γνωστό. Και νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα γιατί το να εστιάσουμε στο διαδίκτυο είναι μεν πιο εύκολο Συγγνώμη, ε, διακόπτει ομιλήτρια, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω έτσι, αλλά αν εξετάσουμε όλες τις περιπτώσεις που συζητούν όλοι πλέον την Ευρώπη, αλλά και εκτός Ευρώπης, για ανθρώπους ε, οι οποίοι ε, ξεφεύγουν ατιμόρυτοι και πράγματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται, νομίζω ότι χάνουμε την αξιοπιστία μας. Πρέπει να συζητήσουμε και τα δύο, τις προτάσεις που έχουμε επιτάπητος, αλλά και τα προβλήματα τα οποία είναι γνωστά σε όλους μας, ε, ξέρουμε ότι υπάρχουν στις χώρες μέλη, σε πολύ μεγάλο βαθμό ε, και ε, σχετίζονται με ε, σεξουαλική κακοποίηση από ε, ιερώμενους. Επίσης, όταν μιλάμε για την πρόληψη, δεν θα πρέπει να μιλάμε μόνο για την τεχνολογία ή δικαστική δράση. Θα πρέπει να αναφερθούμε και στο θέμα του, νομίζω ότι το αναφέρατε εσείς κυρία Σάρμα, της παράδοσης. Και θα ήθελα να προσθέσω της νοοτροπίας μας ως προς τη σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική αγωγή. Διότι σε πολλές περιπτώσεις ένα πρόβλημα είναι πολύ διαστρεβλωμένη και πολύ δυσλειτουργική συμπεριφορά προς τη σεξουαλική μας ε, συμπεριφορά. Ε, και αναγνωρίζω ότι είναι κάτι που δεν συζητάμε πολύ συχνά, αλλά ορισμένες φορές υπάρχουν διαστρεβλωμένες απόψεις για τη σεξουαλικότητα αυτό αποτελεί και τον πυρήνα του προβλήματος και αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αν θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα αυτά. Τέλο, κυρία Πρόεδρε, για το τεχνικό ζήτημα του μπλοκαρίσματο των ιστοσελίδων θα ήθελα να υποστηρίξω τα όσα είπε ο κύριο Μπουταρέλη. Το να μπλοκάρει κάποιο μία ιστοσελίδα δεν είναι απλώ μη αποτελεσματικό, διότι αν ήταν απλώ μη αποτελεσματικό θα έλεγε ένα εντάξει, δεν πιάνει και τι μα πειράζει. Αλλά εγώ δεν είμαι εμπειρογνώμονα, αλλά από τι εξηγήσει που έλαβα, μπλοκάροντας μία ιστοσελίδα, αυτό που κάνουμε ουσιαστικά είναι σαν να ε, κάνουμε ένα τηλεφωνικό κατάλογο για όλες τις άσχημες ιστοσελίδες και σαν να γνωρίζουν όλοι πλέον πού να πάνε να τα βρουν αυτά τα πράγματα. Και νομίζω ότι πετυχαίνουμε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που θέλουμε. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν πάρα πολύ προσεκτικοί με τις λύσεις που αποφασίζουμε να ακολουθήσουμε και να κάνουμε κάτι ώστε να προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο λόγος στην κυρία Ζίπελ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, νομίζω ότι μιλούμε για ένα από τα πιο σημαντικά και τα πιο δύσκολα θέματα και έχουμε μία από, πιο, από τις πιο περίπλοκες και δύσκολες νομοδοτήσεις. Φυσικά όλοι θέλουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταυτόχρονα θέλουμε, έχουμε υποχρέωση να προσέξουμε εάν όλα τα μέτρα τα οποία προτείνονται εδώ στην οδηγία επιτυγχάνουν τον στόχο που θέλουμε να επιτύχουμε. Να μειώσουμε δηλαδή τον αριθμό των κακοποιημένων παιδιών. Και αυτό πρέπει να τύχει ε, βαθιάς μελέτης. Θα συμφωνήσω με αυτά που είπε η κυρία Ινετφέλτ για την κακοποίηση και στον πραγματικό κόσμο μέσα στην οικογένεια, στο οικογενειακό περιβάλλον προς, ε, για, αυτή την, αυτό το πρόβλημα η οδηγία ε, μιλά για την ε, πρόληψη και δίνει πολύ λίγα ως εργαλεία. ήδη ακούστηκαν πολλά σχόλια για την πρόληψη. Τώρα για το θέμα της αύξησης των ποινών. Θα πρέπει να το σκεφτούμε, να δούμε τι θέλουμε να επιτύχουμε καταρχάς με αυτό. Γιατί αν αυξήσουμε τις ποινές, αυτό θα αποτρέψει τους παιδόφιλους που είναι, δεν θα αποτρέψει μάλλον τους παιδόφιλους που είναι, που είναι άρρωστοι. Δεν επιτυχάνουμε τίποτα. Αν τώρα θέλω να πάρω την άλλη ακραία περίπτωση, ότι στα, η, κακοποίηση παιδιών, η κακοποίηση παιδιών έχει να κάνει με εμπόριο ανθρώπων και οργανωμένο έγκλημα, τότε ποιους ε, ε, δράστες θέλω να ε, φυλακίσω αυτόν που βλέπει τις ε, φωτογραφίες, αυτόν που βάζει τις φωτογραφίες στο ίντερνετ ή αυτόν που παίρνει λεφτά από τις φωτογραφίες αυτές. Ελπίζω να προχωρήσουμε τη συζήτηση στον, στο σημείο αυτό. Επίσης, ένα ερώτημα προς την Κομισιόν για το grooming. Γιατί μερικές φορές ε, στις διάφορες μεταφράσεις αυτός ο όρος είναι, ερμηνεύεται διαφορετικά. Τι σημαίνει το grooming. Απ' τη μία υπάρχει αυτό που λέει ότι ε, το grooming σημαίνει έρχομαι σε επαφή με μια web κάμερα με τα παιδιά και τα παιδιά ενθαρρύνονται να, να κάνουν ε, πράγματα τα οποία επίσης διαβιβάζονται μέσω του ίντερνετ ε, και αυτή είναι μία ερμηνεία. Η άλλη ερμηνεία είναι ότι μιλούμε για επαφή με τα παιδιά. Αυτό όμως δεν μπορεί να ποινικοποιηθεί. Αυτό μπορεί μόνο να ποινικοποιηθεί εάν υπάρξει πρόσκληση για σεξουαλική δραστηριότητα σε αυτή την επαφή. Ε, οπότε πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς εννοούμε και τι θέλουμε να ποινικοποιήσουμε. Έχω και άλλες παρατηρήσεις, αλλά εν πάση προς το παρόν ένα τελευταίο σχόλιο τι σημαίνει παιδί, πώς ορίζουμε την ηλικία του παιδιού. Στην οδηγία, όταν μιλούμε για συγκεκριμένες ποινές, συχνά λέμε ότι ε, οι πράσεις ε, ε, ε, εναντίον ενός παιδιού σημαίνει πράξεις ενός, εναντίον ενός ατόμου, ατόμου που δεν έχει φτάσει την ηλικία της, αυτοδιά, της αυτοδιάθεσης. Ε, εντάξει, υπάρχουν διάφορες ερμηνείες ε, ίσως αυτό το θέμα της ε, της ε, ε, αυτό επιδέχεται πολλών ερμηνεών και πολλές φορές λέμε ότι τα παιδιά ε, είναι παιδιά μέχρι την ηλικία των 18. ναι, αλλά και αυτό πάλι είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε. ας δούμε λοιπόν το θέμα της ηλικίας και επίσης τι γίνεται με τις διοκτικές αρχές όταν μπορούν, αν μπορούν να αναγνωρίσουν σε μια ιστοσελίδα αν ένα παιδί είναι 18 ή αν είναι 15. Αυτό είναι σημαντικό για το αν δηλαδή με βάση αυτό μια ιστοσελίδα μπορεί να μπλοκαριστεί ή να κατέβει. Αυτά, Πρόεδρε, από μένα. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Έχουμε πέντε συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο. Θα ήθελα σας παρακαλήσω ο καθένας από τους ευρωβουλευτές να μιλήσει για δύο λεπτά, ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια να προχωρήσουμε και να ακούσουμε τους προσκεκλημένους μας. Αυτός άλλωστε είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε οργανώσει αυτή την ακρόαση. Να ξεκινήσω από τον κύριο Μπρόντς, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κάποιος από τους ομιλητές είπε για τη δυσκολία του να κλείσουν κάποιες ιστοσελίδες. Ε, αν κατάλαβα καλά κάποιες χώρες συνεργάζονται σε αυτό το θέμα. Αναφερθήκαμε επίσης στον σεξουαλικό τουρισμό ή αν ε, προτιμάτε... Ε, σεξουαλικά δεκείμενα που διατράπτονται κατά τη διάρκεια ταξιδιών. Δεν ξέρω αν κάποιες χώρες ε, ε, κοφεύουν ή απλώς είναι ανίκανες να το αντιμετωπίσουν. Όσον αφορά τώρα τις κυρώσεις. Το θέμα της πρόθεσης για αυτά τα αδικήματα, όπως ε, σε όλα τα ε, αδικήματα, μπορεί να είναι προπερασμένο και ανάλογο με τη σοβαρότητα του αδικήματος. Αυτό που δεν μπορεί να είναι πεπερασμένο είναι ε, το γεγονός ε, ότι μπορεί κάποιος να μην ε, ε, δεχτεί την ενοχή του και να, μην, και να βγει νωρίτερα από την φυλακή. Από όσο γνωρίζω, στο Ηνωμένο Βασίλειο όσοι δεν ε, ε, συνεργάζονται δεν σημαίνει απαραίτητα ότι βγαίνουν νωρίτερα. Κατ' εμέ δεν θα έπρεπε να βγαίνουν ποτέ από τη φυλακή. Κάποιο από τους ομιλητές ε, μίλησε εντάχει για το θέμα των αδικημάτων και ορισμένε φορές δεν το γνωρίζει το κοινό. Και οι δημόσιες αρχές δεν λαμβάνουν μέτρα λόγω της ευαισθησίας των τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται οι δράστες. Αυτό επιτρέπει, για παράδειγμα, το grooming ε, κοριτσιών στο Κίθλι, στο Yorkshire, με ελάχιστη κάλυψη από την ε, αστυνομία και με ελάχιστη κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ε, οι οικογένειες ε, των ε, θυμάτων ορισμένες φορές αναφέρονται ως αθώα θύματα και συνήθως είναι. Αλλά ορισμένες φορές κάποια μέλη της οικογένειας παρά το γεγονός ότι δεν έχουν σχέση με το δράστη παριστάνουν ότι δεν γνωρίζουν τίποτα, ενώ δεν τον βοηθούν έτσι να αντιμετωπίσει την ενοχή του, που νομίζω ότι είναι το πρώτο βήμα προ την επανένταξη. Δεν ξέρω πώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, αλλά θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να το αντιμετωπίσουμε. Δεν ξέρω πώ μπορούμε να εντοπίσουμε κάποιον ο οποίο μπαίνει και παρακολουθεί μία ιστοσελίδα παιδική πορνογραφία. Νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνεται κάποιο ε, τέτοιο, αλλά από κάποιε ε, αρχέ ε, σε κάποιε χώρε θεωρείται ότι δεν έχει καμία σχέση ε, με το τι ε, κάνει κάποιος στο διαδίκτυο. Ορισμένες φορές έχουμε κόσμο ο οποίος καταδικάζεται γιατί μπαίνει σε ε, πολιτικές ιστοσελίδες, για παράδειγμα, σε κάποιες χώρες. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε την ίδια σύνδεση. Ευχαριστώ, κύριο Σάλμπρ. Ähm, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας. Μου άρεσαν πάρα πολύ οι παρουσιάσεις. Ε, πραγματικά επικεντρώνονται στα δεδομένα, στα αριθμητικά στοιχεία, ώστε να είναι λίγο πιο ζωντανή η συζήτηση και νομίζω ότι όντως θα πρέπει ε, πάντα να προσπαθούμε να επικεντρωνόμαστε στους αριθμούς και στα γεγονότα και στα δεδομένα γιατί αυτά είναι η πραγματικότητα. Επίσης, από την Κομισιόν ακούστηκε ότι υπάρχουν ε, περισσότερες πληροφορίες με υλικό κακοποίησης παιδιών και πορνογραφικό αν όμως εγώ το έχω καταλάβει καλά, τα τελευταία δύο χρόνια έχει πέσει ο αριθμός αυτών των ιστοσελίδων και αυτό οφείλεται, ε, αυτό το λέει και η έρευνα που έκανε η Κομισιόν και λέει ότι μέσα στην, ε, στην έρευνα αυτή διαπιστώνεται ότι αυτές οι ιστοσελίδες με τέτοιου είδους υλικό τους τελευταίους 6 μήνες, αν διαβάζω εδώ καλά, ε, έχουν μειωθεί κατά 78%. Οι εμπασπιπτώσει έχουν πτωτική τάση. Ε, οπότε μήπως θα μπορούσαμε να το ξεκαθαρίσουμε λιγάκι αυτό. Θέλουμε έτσι λίγο περισσότερες πληροφορίες. Και επίσης, ποιες είναι αυτές οι ιστοσελίδες από αυτές που μπλοκαρίστηκαν, που δεν διαγράφησαν αν έχω καταλάβει καλά, οι περισσότερε από αυτέ τι ιστοσελίδε ή ένα μεγάλο τμήμα του εν πάση περιπτώσει, βρίσκονται στι ΙΠΑ. Ε, Εγώ περιμένω από τι ΙΠΑ συνεργασία στο δικαστικό τομέα. Στενή και άμεση, ώστε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα αυτό. Γιατί μιλούμε για συλλογή δεδομένων, το γνωστό phishing στο ίντερνετ, ε, και βλέπουμε πολλές φορές ε, να κατεβαίνουν ε, ιστοσελίδες που κάνουν αυτή τη συλλογή δεδομένων χωρίς να υπάρχει σύμφωνη γνώμη ε, των πολιτών. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί αυτές μπορούν να κατεβαίνουν και οι άλλες σελίδες με το πορνογραφικό υλικό δεν κατεβαίνουν. Υπάρχει και η σύμβαση για ε, που καταδικάζει την κακοποίηση παιδιών. λοιπόν, έχουμε πολλά δεδομένα στα χέρια μας. και σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή να δούμε αν υπάρχουν και άλλες εναλλακτικέ δυνατότητες ώστε να αντιμετωπίσουμε πιο στεναρά την, ε, το κακό στη ρίζα του. Ή να βοηθήσουμε ας πούμε τα, α, τα θύματα κτλ. Αυτά από μένα πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Βερέιεν. Ναι, Πρόεδρε. Στην Επιτροπή Πολιτισμού ε, εκπονούμε μια ε, γνωμοδότηση για το θέμα αυτό. Το ανέφερε και η συνάδελφος στην αρχή, στα αρχικά του σχόλια. Ένα σημαντικό ζήτημα που δεν συμπεριληφθεί εδώ είναι οι ανταλλαγές από, μεταξύ ομοτήμων peer-to-peer μόνο μέσω των, ανοιχτών προσβα... των ανοιχτά προσβάσιμων ε, στο σελίδων, αλλά και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ χρηστών. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, η καλύτερο, ο καλύτερος δηλαδή συντονισμός και συνεργασία. Ήδη ακούστηκε και για τις σελίδες που κάνουν phishing. μέσα σε δύο ώρες αυτές οι ιστοσελίδες μπορούν να κατέβουν. Οπότε για τις, για τις, για τις σελίδες πορνογραφίας γιατί κρατάει εβδομάδες αυτή η διαδικασία μέχρι να κατέβουν από το ίντερνετ. Γιατί δηλαδή δεν γίνονται πιο άμεσα ε, οι δράσεις αυτές. Ίσως να, υπάρχουν, λοιπόν, να πρέπει να υπάρξουν καλύτερα μέτρα, να υπάρξει καλύτερο συντονισμός, ε, πιο αποτελεσματικά μέτρα έτσι ώστε να χτυπήσουμε το κακό στη, στη ρίζα του. Έχω ακούσει πολλά ενδιαφέροντα σχόλια σήμερα και εδώ νομίζω ότι πρέπει να δούμε πώς μπορούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να δράσουμε, να αντιμετωπίσουμε την παιδική προνογραφία, την κακοποίηση. Ακόμη και τα παιδιά τα οποία ε, δεν έχουν μόνο. Ε, τα παιδιά που δεν την χάνουν κακοποίηση επειδή μπήκαν σε κάποιε σελίδε στο ίντερνετ, αλλά που την χάνουν κακοποίηση και μέσα από το, οικογενειακό του περιβάλλον. Πρέπει ε, τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε, σε σελίδες βοήθειας, σε γραμμές βοήθειας. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να ενισχύσουμε περισσότερο την πρόληψη και να το θέσουμε αυτό ως πολύ βασικό κομμάτι της όλης προσπαθειάς μας. Ευχαριστώ. Grazie. E la parola all'onorevole τώρα. Ja, Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη, Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση δείχνει ότι δεν έχουμε συμπεριλάβει τα πάντα ε, μέσα σε αυτή τη διαδικασία συζήτησης για το ίντερνετ. Εγώ ασχολούμαι χρόνια με την κακοποίηση παιδιών, με την πορνογραφία, με τα όρια που υπάρχουν και, στις, και ακόμη και στις ε, περιοχές μεταξύ ε, Γερμανίας και Τσεχίας και έχουμε πολλά δεδομένα. Υπάρχει ε, πήγουσα ανάγκη δράσης. Ε, βοήθεια προς τα θύματα, πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τα παιδιά, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την πρόληψη ε, αυτό πρέπει να φαίνεται στην, ε, στο κείμενο. Τι γίνεται με τις διαγραφές και, τις, ε, και το μπλοκάρισμα κάποιων ε, ιστοσελίδων ακούσαμε. ποια είναι η εμπειρία που έχουμε, τι γίνεται. Ίσως θα πρέπει πρακτικά να, ενισχύσουμε την όλη συζήτηση αυτή για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόγραμμα. Επίσης, ε, ενίσχυση των ποινών. Εντάξει, ωραία, καλά τα λέμε, αλλά στον τομέα των παιδιών τα, στα παιδιά έχει συνέπεια αυτή η αύξηση των, των ποινών γιατί συνήθως αυξάνεται η βία. Γιατί λέμε αν η ποινή είναι τόσο υψηλή μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο. Μην το υποτιμούμε αυτό. Υπάρχουν πολλά, που, υπάρχουν πολλά δεδομένα που μας λένε να μην αυξήσουμε, να μην οξύνουμε τις ποινές. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τιμωρούμε. Το λόγο έχει η κυρία Βίξτρομ. Εγώ Ήθελα να πω ότι δεν γνωρίζω πολύ καλά την συνάδελφο Σοφία Ιντεβέλτ, αλλά όσον αφορά τα παιδιά και τα σεξουαλικά εγκλήματα, δεν είναι εκτός ε, του σπιτιού που γίνονται όλα αυτά σε κάποιους σκοτεινού δρόμους, αλλά τα περισσότερα, όπως είπε και η Ιντεβέλτ, μέσα στο σπίτι ε, και από ανθρώπους που είναι κοντά στο παιδί, από καθηγητές, ε, μπαμπάδε ε, ή και κληρικούς, παπάδε. Είναι δηλαδή άνθρωποι στους οποίους εμπιστεύονται τα παιδιά και είναι γεγονός ότι στο ίντερνετ διαδίδονται διάφορες ταινίες σε πορνογραφικού περιεχομένου με παιδιά. Αυτά συνεχίζουν να υπάρχουν και αυτά θα συνεχίζουν να ε, παρενοχλούν τα παιδιά για πολλά χρόνια. Είναι ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα αυτή τη στιγμή. Ε, εγώ είμαι υπέρ της ελευθερίας έκφρασης ε, και πρέπει αυτό να είναι ξεκάθαρο. Είναι τόσο σημαντικό οι, διάφορες ε, διάφοροι δημοκρατίες να μπορούν να εργάζονται, να λειτουργούν, να μπορεί ο καθένας άνθρωπος να γράφει και να εκφράζεται. Και αυτό θα πρέπει να ισχύει και στο ίντερνετ. Αλλά υπάρχουν και όρια όσον αφορά την ατοπική ελευθερία από τη στιγμή που ε, θίγει την, ε, τα παιδιά. γιατί αυτό τους αφαιρεί το δικαίωμα στην ακαιρεότητα και ε, καταπατά δηλαδή τα όρια της ελευθερίας των ίδιων των παιδιών. Η παιδική πορνογραφία δεν σημαίνει μόνο το, την παραβίαση ενός ορίου ελευθερίας έκφρασης. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το μπλοκάρισμα ως ένα μέσο υπεράσπισης των δικαιωμάτων των παιδιών. Το καλύτερο είναι να μπορούσαμε να διαγράψουμε αυτά τα site στην πηγή, στην αρχή. Και αν δεν γίνεται κάτι τέτοιο, τότε να χρησιμοποιήσουμε το μπλοκάρισμα. Βεβαίω και να επικρατεί δημοκρατία και ελευθερία έκφραση στο ίντερνετ, αλλά δεν επιτρέπονται όλα. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να είναι αποδεκτό. Ο κύριος Μπουταρέλη ακριβώς περί αυτού μίλησε ότι θα πρέπει να θυμόμαστε ότι θα χρειαστεί να καταλήξουμε σε μια ισορροπία. Είναι δυνατόν να προστατεύσουμε την ακυρεότητα των παιδιών χωρίς να θέσουμε υπό αμφισβήτηση την ελευθερία στο ίντερνετ. Θα πρέπει δηλαδή πάντοτε να έχουμε υπόψη μας το εξή, ε, καθώς εργαζόμαστε πάνω σε αυτό το θέμα. Μιλάμε για σοβαρότατα εγκλήματα, τα οποία διαπράττονται στο ίντερνετ, αλλά διαπράττονται και πολύ πιο κοντά στην ε, αληθινή ζωή των παιδιών. Eh, Σας ευχαριστώ και τώρα το λόγο ε, για την τελευταία παρέμβαση έχει η κυρία Μπλίνκη Τσούτη. Σας ευχαριστώ. Οι βάσει δεδομένων πορνογραφία βασικά έχουν έδρα τη ΣΥΠΑ, την Αυστραλία και κάποιε ευρωπαϊκέ χώρε. Και όπω είπε και η επίτροπο Μάλμστρομ σε προηγούμενη τη παρέμβαση, συνεχίζονται συζητήσει και διαπραγματεύσει με την ΣΥΠΑ και τη Ρωσία για να μπλοκαριστούν αυτές, αυτοί οι σερβερ. Υπάρχουν όμω κάποια κατημέλη που δεν κάνουν τίποτα. Δεν νομίζετε ότι θα ήταν πιο αποτελεσματική η δράση το να υπάρξει μία διεθνής δεσμευτική συμφωνία νομικά δεσμευτική συμφωνία γιατί νομίζω πως απλώς οι διμερείς συμφωνίες δεν πρόκειται να λειτουργήσουν Επίσης πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί πιο σοβαρή ποινική ευθύνη για αυτά τα αδικήματα και συμφωνώ με την κυρία Αντζελίλη που είπε ότι θα πρέπει να έχουμε μια γενική πολιτική στρατηγική μάλλον πρόληψη. Μπορούμε να έχουμε τέτοια στρατηγική πρόληψη αν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει κάποια, δεν, δεν έχουμε στοιχεία που να μας δείχνουν πόσο ε, διαδεδομένο είναι αυτό το φαινόμενο. ας κουνηθούν τα κρατημέλη, ας αρχίσουν να συλλέγουν τέτοιου είδου στοιχεία. Αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε την σεξουαλική παρενόχληση των παιδιών και την παιδική πορνογραφία, θα πρέπει να κάνουμε συντονισμένες προσπάθειες. Γι' αυτό και πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να ε, ε, ε, κατανείμουμε ευθύνε, να πούμε δηλαδή ότι τα κράτη-μέλη θα είναι υπεύθυνα για τη θέσπιση των μήνυμων ποινών ή των μήνυμων κυρώσεων για τέτοιου είδου παραπτώματα. Δεν νομίζω πω αυτή είναι η ζωστή προσέγγιση. Αν θέλουμε να έχουμε πραγματικά αποτελέσματα, θα πρέπει όλοι να συνεργαστούμε. Και γι' αυτό και οι μήνυμων ποινέ θα πρέπει να θεσπίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και μια τελευταία παρατήρηση. Έχουμε προσωπικό το οποίο να είναι κατάλληλα καταρτισμένο ώστε να κάνετε τέτοιου είδους προγράμματα. Δεν το έχουμε αναφέρει ακόμα αυτό, αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως η κοινωνική λειτουργή, η εκπαιδευτική, όλοι θα πρέπει να έχουν ιδιαίτερη κατάρτιση, ώστε να μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν τα παιδιά να μιλήσουν για τέτοιου είδους ε, παρενοχλήσεις. Δεν πρέπει αυτό να το ξεχάσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω καταρχάς ε, τους ομιλητές ε, για αυτό το πάνελ εργασίας. Ε, για άλλη μια φορά να σας ζητήσω να στείλετε στη γραμματεία της ε, ε, Επιτροπής μας την παρέμβασή σας, ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε με το βέλτιστο δυνατό τρόπο τις παρατηρήσεις που μας έκαναν σήμερα. Και να ζητήσω τώρα από τον κύριο Λορέλ και τον κύριο Έρτινγκ εκ μέρους της Eurojust και της Europol να έρθουν εδώ στο Προεδρείο. Ευχαριστώ πολύ.

Okay. Ehm, λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα τις εργασίες μας και να δώσουμε αμέσως το λόγο στον κύριο Λαουρέλ ε, Eurojust. Πρέγω. Τον εκπρόσωπο της Eurojust. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Είμαι μέλος της Σουηδίας ε, για το Eurojust. Αυτό βέβαια δεν λέει τίποτα. Είμαι εισαγγελέα και άσω μια πιο επιχειρησιακή άποψη για την οδηγία και θα σας δώσω και ένα παράδειγμα από την πραγματικότητα. Eurojust is the judicial cooperation η Eurojust είναι ο ευρωπαϊκός οργανισμός για την Ευρώπη, το δικαστικό δίκτυο και εμείς συντονίζουμε τις δράσεις μας ε, για θέματα έρευνας και εισαγγελικών ε, διώξεων. Ε, ασχολούμαστε με σοβαρά διαμεθοριακά αδικήματα, κυρίως οργανωμένο έγκλημα. Επίσης, διευκολύνουμε τη συνεργασία μεταξύ των δικαστικών αρχών στα κράτη-μέλη και επίσης με τρίτες χώρες. Και είμαστε και κέντρο εμπειρογνωμοσύνης για διεθνή δικαστικά θέματα, κυρίως σε θέματα συνεργασίας μεταξύ χωρών. Κάποια σχόλια για το σχέδιο οδηγίας. Θα σας αναφέρω κάποια υπέρ και κάποια κατά. Το θετικό είναι ότι σοβαρές μορφές σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης που δεν καλύπτονται από την παρούσα ευρωπαϊκή νομοθεσία πλέον τιμωρούνται. Θα επικεντρωθώ στα τμήματα της οδηγίας που ενδιαφέρουν περισσότερο τις βασικές εργασίες της Eurojust. Αυτό που είναι θετικό είναι το γεγονός ότι η νέα οδηγία θα τιμωρεί νέα φαινόμενα στο ε, περιβάλλον της πληροφορικής. Θα υπάρχει καλύτερος ε, ε συντονισμός σε θέματα σεξουαλικών ειδικημάτων κατά παιδιών και ένα καλύτερο νομικό πλαίσιο. Και θεωρούμε ότι είναι θετικό το γεγονός ότι αναφερόμαστε ε, και στην ε, απόφαση πλαίσιο για την επίλυση διαφορών ε, σε νομικές διαδικασίες και ο ρόλος της Eurojust περιγράφεται ακριβώς εκεί, στο νομικό πλαίσιο. Θέματα δικαιοδοσίας για αυτή τη μορφή τα δικήματα μπορεί να είναι πάρα πολύ σοβαρά. Uh, Θα ήθελα να συμφωνήσω με την κυρία Σάρμα ότι όροι όπως ο σεξουαλικός τουρισμός και η παιδική πορνογραφία είναι μάλλον αδόκιμοι. Θα ήθελα να προτείνω, όπως είπε και η κυρία Σάρμα, να έχουμε ε, παραβάτες ε, σεξουαλικών αδικημάτων ε, κατά τη διάρκεια ταξιδίων και εικόνες κατά κακοποίησης παιδιών. Οποιαδήποτε εικόνα παιδιού σε κάποια σεξουαλική συμπεριφορά η οποία βρίσκεται στην οδηγία, περιγράφεται εξορισμού στην οδηγία, είναι περιγραφή εικόνας αδικήματος. Δεν θα πρέπει να γίνεται εδώ σύγχυση μεταξύ των νομικών περιγραφών, της πορνογραφίας δηλαδή, και της παιδικής πορνογραφίας με την παράνομη περιγραφή αυτού του αδικήματος. Δεν είναι μια άλλη μορφή πορνογραφίας, πρόκειται για μια απεικόνηση αδικήματος. Εγκλήματος. Υπάρχουν νέες δυνατότητες όπως αναφέρθηκε να χρησιμοποιήσουμε νέα ερευνητικά ε, μέσα και μία έρευνα δεν θα εξαρτάται ε, μόνο από μία αναφορά ή μία κατηγορία εκ μέρους του θύματος ή εκ μέρους της οικογένειας του θύματος επειδή ακριβώ υπάρχουν σαφείς ορισμοί για τα εγκλήματα που διαπράττονται, ε, είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά όπως σα είπα και στην αρχή, θα πρέπει κάποιοι όροι να επανεξεταστούν. Ένα από τα σημαντικά θέματα είναι η εκτιτεμένη ε, ε, δικαιοδοσία, η εξοεδαφικότητα. Όχι μόνο η δυνατότητα να ε, δικαστούν ε, και να διωχθούν ε, ταξιδιώτες οι οποίοι ε, διαπράττουν σεξουαλικά δικήματα, αλλά οποιαδήποτε άλλα δικήματα διαπράχθηκαν εκτός ε, εδαφικής και οδησίας να διώκονται εξοεδαφικά. Δεν θα σταθώ σε θέματα όπως είναι η αφαίρεση υλικού από ιστοσελίδες, αλλά θα ήθελα απλώς να σας υπενθυμίσω εδώ ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα δικαιοδοσίας. Είναι εύκολα τα πράγματα όταν έχουμε ένα σερβερ σε ένα κράτο ή στι Ηνωμένε Πολιτείε, διότι εκεί υπάρχει καλή συνεργασία με τι Ηνωμένε Πολιτείε και μπορεί να λυθεί το θέμα, αλλά θα μπορεί να υπάρξει πρόβλημα εάν ο σερβερ βρίσκεται σε μια χώρα με την οποία δεν έχουμε συνεργασία. Αν αφαιρεθεί υλικό, ε, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία ώστε να μπορούμε να το κάνουμε στην επικράτεια άλλου, άλλου, Τώρα, κάποια στατιστικά στοιχεία. Έχουμε στατιστικά στοιχεία από τις υποθέσεις με τις οποίες έχει ασχοληθεί η Eurojust. Όπως βλέπετε δεν είναι πάρα πολλές αυτές οι υποθέσεις, αλλά εμείς ε, ασχολούμαστε με σοβαρά εγκλήματα. Ε, πολλές φορές υπάρχει εμπλοκή και πολλών κρατών μελών ε, ή και τρίτων ε, χωρών. Επομένως δεν μιλάμε για συνήθι αδικήματα σεξουαλική κακοποίησης που διαπιστώνονται σε ένα κράτο μέλος. Πρόκειται για περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν πολλές χώρες μέλη συχνά. Το 30% των περιπτώσεων είναι περιπτώσεις σεξουαλικής ε, κακοποίησης, ε, συμπεριλαμβανομένων διασμών και σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Ένα 10% είναι ε, αυτά τα οποία αποκαλούμε παιδική πορνογραφία, 14% εγκλήματα κατά της ε, ζωής και της προσωπικής ελευθερίας και περιλαμβάνουν σε αυτά τα στατιστικά στοιχεία 9 φόνους και μία ανθρωποκτονία. Θα περιγράψω εν συντομία μία υπόθεση που νομίζω είναι ένα καλό παράδειγμα ε, για να αντιληφθείτε τι ακριβώς υποθέσεις εξετάζουμε εμείς ε, στην Eurojust πρόκειται για την υπόθεση του χαμένου αγοριού. Εδώ είχαμε αρκετέ χώρες ε, οι οποίε ενεπλάκησαν και πρόκειται για εξάρθρωση ενός παγκόσμιου ε, δικτύου παιδοφιλίας. Η υπόθεση ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2007. Είχαμε μία αίτηση αμοιβαία ε, δικαστικής συνδρομής από Νορβηγία στην Ιταλία. Εστάλθηκε αυτή η αίτηση μέσω Eurojust γιατί συνήθως η εφαρμογή του νόμου και τα δικαστικά δίκτυα που χρησιμοποιούνταν συνήθως δεν ε, λειτουργήσαν. Επομένως η Νορβηγία ζήτησε τη συνδρομή της Eurojust. Η Νορβηγία έχει μία συμφωνία συνεργασίας ε, με τη Eurojust και, ένας, και υπάρχει και εισαγγελέα ε, σύνδεσμο ε, της Νορβηγία, ο οποίος εργάζεται στη Eurojust. Ε, έχουμε πολύ σοβαρά σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών και έχουμε χιλιάδες φωτογραφίες σεξουαλικής κακοποίησης και πάρα πολλές ταινίες. Υπήρξε ένα τεράστιο δίκτυο το οποίο λειτουργούσε ως επιχείρηση και παρήγαγε και διένυμε ε, υλικό σεξουαλικής κακοποίησης. Αλλά τα μέλη του δικτύου αυτού ε, κακοποιούσαν παιδιά ε, και τα ίδια. Χρησιμοποίησαν φυσικά το διαδίκτυο. Το δίκτυο βασιζόταν σε ελεύθερο λογισμικό αλλά ε, οι, υπηρεσί, οι σερβερ άλλαζαν συνεχώς και είχαν τεχνολογικά ε, προηγμένα πρωτόκολλα ασφαλείας. Ε, βλέπετε εδώ στις εικόνες ότι είχαμε έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Βέλγιο, στη Βραζιλία, στον Καναδά, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στο Μεξικό, στις κάτω χώρες, στη Νέα Ζηλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. 35 μέλη ε, εντοπίστηκαν και πάρα πολλά θύματα παγκοσμίως. η Eurojust διευκόλυνε τη συνεργασία μεταξύ των χωρών αυτών και έκανε και πέντε συντονιστικές συνεδριάσεις, τις οποία στις ανακριτές και εισαγγελείς στις ε, λόγω χώρες συναντήθηκαν, αντάλλαξαν πληροφορίες, αντάλλαξαν και αιτήσει αμοιβαία συνδρομής και ε, συντόνισαν τις δράσεις τους. Είχαμε μία καταδίκη στην Νορβηγία, 10 χρόνια ε, κράτηση και η υπόθεση συνεχίζεται διότι έχει προσφύγει στο εφετείο ο δράστης. Είχαμε χιλιάδες ε, ε, πορνογραφικές εικόνες οι οποίες κατασχέθηκαν και εντοπίστηκαν και 17 θύματα. Είχαμε θύματα από την Ορβηγία, τη Ρουμανία και τη Βραζιλία. Στην Ιταλία συνελήφθη ένας από τους δράστες. Είχαμε κατάσχεση άνω του ενός εκατομμυρίων φωτογραφιών. Επτά θύματα και δύο ενδιάμεση εντοπίστηκαν στη Ρουμανία. Στη Ρουμανία είχαμε 8 άτομα που έκαναν στρατολόγηση ε, και τους βρήκαμε, ε, βρήκαμε και 27 θύματα μέσω φωτογραφιών. Στις Ηνωμένε Πολιτείες 15 μέλη εντοπίστηκαν 14 εξ αυτών ε, βρίσκονται υποκράτηση και κατά πάσα πιθανότητα θα λάβουν ποινή φυλάκισης ε, τουλάχιστον 20 ετών. Είχαμε 25 θύματα και 7 τεραμπάιτ ε, πορνογραφικού υλικού το οποίο κατασχέθηκε. Το 1 τεραμπάιτ είναι 1 εκατομμύριο μεγαμπάιτ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρόκειται για πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα υλικού. Δεν έχω ξανακούσει αντίστοιχη κατάσχεση υλικού ε, στο παρελθόν. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαμε ένα δράστη, στη Γαλλία είχαμε σύλληψη ενό ατόμου, στην Βραζιλία τέσσερα άτομα και στο Βέλγιο εντοπίστηκε και συνελήφθη ένα άτομο. would have been impossible to coordinate these actions επειδή ακριβώς ε, είχαμε εμπλοκή τόσων πολλών κρατών μελών, θα ήταν αδύνατο να ε, συντονιστούν όλες αυτές οι δράσεις αν δεν υπήρχε κάποιος διεθνής οργανισμός όπως η Eurojust. Η Eurojust είναι πλάκη διότι οι ε, συνήθεις διάβλοι δεν ε, είχαν αποτέλεσμα και συντόνισε τις δράσεις μέσω συνεδριάσεων και στη Χάγη και στα διάφορα κράτη-μέλη προκειμένου οι ερευνητές και ανακριτές ε, να συναντηθούν και να συντονιστούν. Να σας ε, δείξω ένα παράδειγμα εδώ στην οθόνη. Ένας εισαγγελέας από τις Ηνωμένε Πολιτείες μία συγγνώμη, έφερε προσωπικά ε, στοιχεία και ξεκίνησε την έρευνα στις Ηνωμένε Πολιτείε και βλέπετε εδώ το αποτέλεσμα, συνελήφθησαν 15 άτομα και οι 14 εξ αυτών βρίσκονται υποκράτηση. Πρόκειται για μια πολύ επιτυχή συνεργασία. Ξεκίνησε το 2007 και ακόμα δεν έχουμε δει όλα τα αποτελέσματα, ε, αλλά μπορείτε να δείτε κάποια εξ αυτών εδώ στην διαφάνεια. Αυτές είναι και οι πληροφορίες ε, για το πώς μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. Γι' αυτό θα ήθελα να σας συζητήσω να μας τη στείλετε και να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Έρτινγκ, εκπρόσωπο της Europol. Παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν ευχαριστώ την Επιτροπή σας που οργάνωσε αυτή την πολύ σημαντική ακρόαση. Η Europol φυσικά καλωσορίζει τις δραστηριότητε του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, των κρατών μελών της Κομισιόν προς αυτό το σκοπό το 2009 ήδη, κατά τη διάρκεια των αρχικών φάσεων της εκπόνησης αυτού του προγράμματος, η, προ, η, Europol είχε κάνει μια συνάντηση με εμπειρογνώμονες. Μιλούμε για ε, εμπορία, σεξουαλική εκμετάλλευση, ε, οι οποίες έχουν τεθεί ως προτεραιότητες για την Europol και παρόλο που εγώ είμαι 30 χρόνια στο αστυνομικό σώμα, ακόμη σοκάρομαι όταν πηγαίνω στη μονάδα για, την, για σεξουαλική εκμετάλλευση και μου δείχνουν παραδείγματα νέων θηριωδιών που γίνονται εναντίον των παιδιών. Η Europol έχει συντονίσει και συμμετάσχει σε πολλέ επιχειρήσει στα κράτη-μέλη. Το, στο τέλη του 2010, φέτος, έχουμε υποστηρίξει πάνω από 30 διεθνείς υποθέσεις που έχουν να κάνουν με ποινικά, ε, με εγκληματικότητα, με ε, ε, και σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και διαβίβαση του υλικού. Έχουν βρεθεί πάνω από 2.000 υποπτοί και επίσης έχει βρεθεί και ένας μεγάλος αριθμός θυμάτων. Έχουμε πάρα πολλά εργαλεία και μέσα που από κοινού χρησιμοποιούμε με τα κράτη-μέλη ώστε να, να βρούμε ποιοι είναι οι πιο στιγνοί εγκληματίε στο... στην Ευρώπη. Έχουμε βρει περίπου 40.000 περιπτώσει ε, διασυνοριακών ερευνών που μας δίνουν έτσι μια γενική εικόνα του τι γίνεται σε ποινικό επίπεδο στην Ευρώπη. Τώρα, για την πρόταση που υπάρχει επιτάπητος. Να σα πω ποιοι είναι οι τομεί που μας ενδιαφέρουν εμά περισσότερο. Σε ό,τι αφορά το, τους ορισμούς, την παιδική πορνογραφία, το παιδί, την ε, εκπόρνευση, ε, όντως δεν είναι σαφής ο ορισμός τους. Ε, προφανώς πρέπει να υπάρξει καλύτερος ορισμός που να είναι και συνεκτικός με τα διεθνή εργαλεία που υπάρχουν. Μια τέτοια ε, γενική συνολική ε, προσέγγιση θα βοηθήσει και θα ενισχύσει τις ε, προσπάθειε που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της, ε, του προβλήματο αυτού. Τώρα για τα άρθρα 3-7 7 που μιλούμε για την εκμετάλλευση των παιδιών, τη σεξουαλική κακοποίηση που δεν καλύπτονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία πλέον θα ποινικοποιούνται. Η Europol καλωσορίζει την εισαγωγή μια νέα διάταξη που περιλαμβάνεται στο άρθρο 5 και που ποινικοποιεί την παράνομη δραστηριότητα νομικός, νομίμως αποκτηθέντο υλικού που έχει να κάνει με παιδική πορνογραφία. Η Europol ε, και η εμπειρία της δείχνει ότι οι χρήστες του ίντερνετ που κατεβάζουν υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης είναι και παραγωγή ή οι διανομής αυτού του παράνομου προϊόντου, υλικού. Ε, η η διανομης αυτου του παρανομου λοιπόν και η διανομή αυτού του υλικού ε, βρίσκεται μετά την έρευνα στις εγκαταστάσεις. γιατί πολλές φορές οι δράστες ε, ε, βλέπουν πολλές, ε, κάνουν έτσι μια, ένα ξεσκαρτάρισμα των ιστοσελίδων χωρίς όμως αναγκαστικά να καταλήγουν ή να κατεβάζουν σε κάποιο, κάποιο υλικό. Παρ' όλα αυτά αυτή η πράξη πια ποινικοποιείται. Επίσης, και είναι πολύ σημαντικό, Υπάρχει ένας νέος, ένα νέο modus operandi που μας επιτρέπει να βρίσκουμε ε, ακόμη και ε, από, ε, υλικό που έχει αποθηκευθεί σε δίσκους εκτός των κομπιούτερ των χρηστών ή σε web hotels που υπάρχουν πλέον ή σε άλλους χώρους στο διαδίκτυο. Άρθρο 6. Νέοι, νέοι τρόποι εκμετάλλευσης και κακοποίησης που διευκολύνονται από το ίντερνετ ποινικοποιούνται. Ε, online grooming για παράδειγμα. Η Europol υποστηρίζει την ε, διάταξη αυτή γιατί το online grooming είναι πραγματικότητα, συμβαίνει. Μάλιστα, ε, όχι μόνο οι έφηβοι αλλά και μικρότερα παιδιά έρχονται σε επαφή με παιδόφιλους για οποιαδήποτε... Για, δραστηριότητες κακοποίησης. Είναι πάρα πολύ απλό άλλωστε. Μια σύνδεση στο ίντερνετ χρειάζεται και η Europol μέσω των κοινωνικών ιστοσελίδων ε, προσπαθεί να ενισχύσει την ε, συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα ε, ώστε να, μπορέσουν, να, μπορέσει να περιοριστεί το φαινόμενο αυτό. Δηλαδή να υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος των παιδιών, ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να καταχωρούνται ή να χρησιμοποιούν σελίδες που αφορούν μόνο είτε εφήβους είτε ενηλίκους. Επίσης θα υπάρξει μια νέα διάταξη για τη βοήθεια σε έρευνες και να μπορούν να, οι ένοχοι να έρχονται ενώπιον του δικαστηρίου και να τιμωρούνται. Ε, το άρθρο 40 τώρα. Η Europol έχει αντιμετωπίσει πολλέ υποθέσει σε κάποια κρατημέλη, όπου το θύμα ε, αναγνωρίστηκε μετά από πολλά χρόνια και έχει ήδη ενηλικιωθεί. Σε κάποιες περιπτώσεις ε, ο ε, παιδεραστής επίσης ε, αναγνωρίστηκε μετά από κάποια χρόνια αν και το θύμα μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να μην ήθελε να τον ασκήσει δίωξη γιατί έχουν περάσει, έχει περάσει πάρα πολύ καιρό από τότε. Οπότε σε τέτοιε περιπτώσει ο παιδόφιλο αναγνωρίζεται μεν, δεν κατηγορείται δε. Φυσικά αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ξαναεπιχειρήσει να κάνει κάτι τέτοιο με άλλα παιδιά. Άρθρο 14. Η Europol ε, θεωρεί ότι, είναι, ε, ότι αξίζει τον κόπο να προσθεθούν και άλλα μέτρα ώστε να αναγνωρίζονται τα θύματα τη παιδική πορνογραφία μέσω τη χρήση των τεχνολογιών, όπω α πούμε η ανάλυση εικόνων. Από επιχειρησιακή πλευρά, αυτή η έρευνα και αυτή η τεχνική όντω έχει αποδειχτεί πολύ χρήσιμη για να, και επιτυχάνει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Η αναγνώριση και η δυνατότητα τη διάσωση του παιδιού είναι πολύ σημαντικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά το άρθρο 16 ε, για την αδικαιοδοσία ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι ε, εγκληματίες θα έρχονται ενώπιον του δικαστηρίου. Είναι σημαντικό οι παιδεραστές να έχουμε υπόψη μας ότι ε, μετακινούνται συνέχεια ή ταξιδεύουν από χώρα σε χώρα ώστε να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα παιδιά επιτόπου. Οι ε, εγκληματίες αυτοί δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε νομοθεσία και ακριβώ επειδή θέλουν να αποφύγουν τις ποινικέ διώξεις στη χώρα καταγωγή τους μεταφέρονται από χώρα σε χώρα. Η Europol στο παρελθόν έχει αντιμετωπίσει πολλές τέτοιες περιπτώσεις όπου ο επαγγελματίας αυτός ε, ταξίδευε από χώρα σε χώρα πολύ συχνά. Η διάταξη λοιπόν που υπάρχει στο 16 πάει προς σωστή κατεύθυνση γιατί ακριβώ καλύπτει τα κενά που υπήρχαν στην νομοθεσία μέχρι στιγμή. Η Europol θα ξεκινήσει μια πρωτοβουλία ώστε να ε, βρει αυτούς τους εγκληματίες ε, από κοινού με, τους, με τις ποινικές αρχές των κρατών μελών. Ένα τελευταίο σχόλιο και το άρθρο 19α και 21 για τα επιπλέον μέτρα που πρέπει να αποτρέψουν τον σεξουαλικό τουρισμό και να χρησιμοποιηθεί ο εθνικός, ε, ο εθνικός μηχανισμός για να μπλοκαριστούν ιστοσελίδες ε, που βρίσκονται εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Europol υποστηρίζει ότι η ε, αντιμετώπιση του προβλήματος αυτό χρειάζεται και μια πολυσχηδή προσέγγιση γιατί ακριβώς λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχει αυτό το ιδιαίτερο έγκλημα. Επίσης, συνεργασία ιδιωτικού και δημοσίου τομέα που μπορεί να μας, ε, να μας ε, ε, προειδεάσει για κάποιε ιστοσελίδε που επισκέπτονται συγκεκριμένα άτομα ε, ώστε να προλάβουμε ε, δικήματα. Επίση, ε, η Europol έχει υποστηρίξει την δημιουργία μια τεχνολογία φιλτραρίσματο σε κάποια κράτη-μέλη. Με την τεχνολογία αυτή εφαρμόζουμε, εφαρμόζουμε μέσω των providers, των παρόχων, το φιλτράρισμα των διαφόρων ιστοσελίδων. Παρόλο που το, μπλο, το μπλοκάρισμα είναι η τελευταία λύση για την αντιμετώπιση των ιστοσελίδων αυτών, θεωρείται ω αρκετά ικανοποιητικό μέτρο για την αντιμετώπιση του προβλήματο ε, μέσα στο ίντερνετ. Τούτου λεχθέντος, ε, το τελικό σχέδιο κειμένου θεωρούμε ότι αποτελεί μια σταθερή βάση για να υπάρξει μια συνεκτική ε, νομοθεσία για την αντιμετώπιση του σεξουαλικού εγκλήματο. Η Europol θεωρεί ότι είναι πολύ θετική η πρόταση που έχει υποβάλει η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ehm, eh, Σα ευχαριστώ. Πριν αρχίσουμε τη συζήτηση θα δώσω το λόγο στη, καταρχήν στην Ρεζίνα Γιάννη Στότερ που αντιπροσωπεύει το, το Συμβούλιο της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Ένα στα πέντε παιδιά πέφτουν θύματα, πέφτει θύμα σε μορφής, κάποιες μορφής ε, βίας, παρενόχλησης ή κακοποίησης. Το 80% αυτών των παιδιών πέφτουν θύματα αυτού του είδους βία στον κύκλο εμπιστοσύνη τους, όπως αποκαλείται. Δηλαδή, μέσα στην οικογένεια ή σε ε, ιδρύματα είτε από φίλους γνωστούς. Ε, αυτό πρέπει να το φροντίσουμε να σταματήσει. Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που συγκέντρωσε πολλούς εμπειρογνώμονες αλλά και υπαλλήλους ψηλού επίπεδου για αυτό το είδος την ακρόαση. Είναι πλέον καιρός να δράσουμε και πιστεύω πως αυτή η ακρόαση θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε. Στα 10 λεπτά που έχω στη διάθεσή μου θα σας παρουσιάσω τις βασικές διαφορές ανάμεσα στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών από την σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση και το σχέδιο οδηγίας ε, που συζητάμε σήμερα. Θα σας δώσω και την τελευταία ενημέρωση για τη μελλοντική εκστρατεία του Συμβουλίου της Ευρώπης για να σταματήσει η σεξουαλική βία κατά των παιδιών. Ε, συνοδεύομαι από μία συνάδελφο από το τμήμα ποινικού δικαιού του Συμβουλίου της Ευρώπης που θα μπορέσει να απαντήσει σε τεχνικής φύσης ερωτήσεις όσον αφορά τη σύμβαση ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτή έχει υπογραφεί ε, από 39 κράτη-μέλη μέχρι στιγμής. 8 επικυρώσεις είναι υπό εξέλιξη. Αλβανία, Δανία, Ελλάδα, Μάλτα, κάτω χώρες, Άγιος Μαρίνος, Σερβία και Ισπανία. Περισσότερες επικυρώσεις αναμένονται το πρόβλημα της σεξουαλικής βίας κατά των ε, παιδιών ε, είναι παγκόσμιο και είναι ανοιχτή η σύμβασή μας για υπογραφή και επικύρωση και από μη κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και έχει εκφραστεί ενδιαφέρον εκτός Ευρώπης, ιδιαίτερα από αυτούς που συμμετείχαν κατά τη διάρκεια της σύνταξης. ΗΠΑ, Ιαπωνία, Καναδάς, Μεξικό. Η σύμβαση μπορεί επίσης να επικυρωθεί από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θα ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο. Η σύμβαση είναι δυναμική με την έννοια ότι έχει στόχο να συμβαδίσει με την εξέλιξη των εγκλημάτων και τον τρόπο αντιμετώπιση του Εισάγονται δεσμευτικέ διαδικασίε που θα παρακολουθήσουν τη συμμόρφωση, τη διευκόλυνση κοινή ερμηνεία και εντοπισμό καλών πρακτικών δεν είναι νομικό μέσο που ασχολείται μόνο με το ποινικό δίκαιο. Θέλει να εισάγει νέα μέτρα, ε, περαιτέρω μέτρα για τις διεθνείς συμβάσεις και την προστασία των θυμάτων. Είναι μια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει το καλό παράδειγμα. Η παιδεία και η ενημέρωση είναι σημαντικό κλειδί. Τα άρθρα 5 με 10 έχουν στόχο την αύξηση της ενημέρωσης των ίδιων των παιδιών, των όσων εργάζονται με τα παιδιά και με το ευρύτερο κοινό εκτός από την εφαρμογή των μέτρων ε, παρέμβασης, κατοικής παρέμβασης σε σχέση με τους δράστες, ε, θέλουμε να υπάρξει συνεργασία για τον εντοπισμό και την δίωξή τους. Η Σύμβαση έχει τέσσερις κύριους στόχους να παρεμποδίσει και να καταπολεμήσει την σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση των παιδιών, να προστατέψει τα δικαιώματα των θυμάτων, να προωθήσει την εθνική και τη διεθνή συνεργασία κατά τέτοιου είδου εκμετάλλευση και να ενθαρρύνει την εφαρμογή μέσω τη δημιουργία ειδικών ε, μηχανισμών εποπτεία, ώστε να διασφαλιστεί ότι το σύστημα αυτό εφαρμόζεται και να ενθαρρύνει τη συνεργασία ανάμεσα στα 47 κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η σύμβαση δεν ορίζει νομικές ε, έννοιες εξαιρετικά περιοριστικά και δεν υπάρχει συγκεκριμένο ορισμός για τη σεξουαλική δραστηριότητα ή για την σεξουαλική συμπεριφορά ή την πορνογραφική ε, συμπεριφορά. Αυτό επιτρέπει στα κράτη-μέλη να τα ορίσουν όλα αυτά στο πλαίσιο των δικών τους νομικών ε, συστημάτων. Και η ηλικία σεξουαλικής συγκατάθεσης δεν ορίζεται επίσης γιατί είναι σαφές ότι η νομοθεσία των κρατών μελών ποικίλει από τα 13 μέχρι τα 17 έτη ως όριο ηλικία συγκατάθεσης. 47 λοιπόν κράτη-μέλη τα οποία μπορούν να συμμορφωθούν ανάλογα με το πώς θεωρούν ε, ότι πρέπει και ανάλογα με τις ε, περιστάσεις κάθε φορά. Τα νομικά συστήματα των κρατών μελών ε, δεν είναι αρκετά εναρμονισμένα γιατί ε, δεν έχουν εναρμονιστεί στο βαθμό που έχουν εναρμονιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή είναι ε, μια ακόμα ευκαιρία για την Ένωση. Παρομοίω, οι ποινέ ε, δεν είναι προκαθορισμένε ενώ θα έπρεπε να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και ε, πιστικές. Ε, το Συμβούλιο της Ευρώπης γνωρίζει πως τα κράτη-μέλη θέλουν να διατηρήσουν τον έλεγχο αυτής της πτυχής της νομοθετικής διαδικασίας και γνωρίζει πως σημαντικές διαφορές μπορεί να υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Εμεί θεωρούμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το σχέδιο τη Οδηγία δεν θα περιορίσει το πεδίο εφαρμογή της σύμβαση και ότι οι διατάξει θα είναι ε, εφαρμοστές, ε, αναλογικές και αποτρεπτικές. Υπάρχουν δύο βασικές διαφορές ωστόσο ανάμεσα στη σύμβαση και το σχέδιο οδηγία. Οι ορισμοί και η πρόταση της Ένωσης να εφαρμόσει και τεχνολογία μπλοκαρίσματος ή διαγραφής σε site, στα site που περιλαμβάνουν τέτοιο υλικό. Έχουμε το στόχο του μέσου καθώς και το λεπτομερή ορισμό των ε, διαφόρων όρων και όλοι συμφωνούμε ότι βασικός στόχος είναι η προστασία των παιδιών και η τιμωρία της ε, σεξουαλικής ε, παρενόχλησης και κακοποίησης των παιδιών. Ωστόσο, οι διαφορές αυτές θα πρέπει να σημειωθούν. Η σύμβαση έχει βασικό στόχο την πρόληψη, την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων, την προώθηση εθνικής και διεθνούς συνεργασίας και τη δημιουργία ενός ε, μηχανισμού παρακολούθησης για την εφαρμογή της σύμβασης. Αντίθετα, το σχέδιο οδηγίας ε, έχει πιο περιορισμένους στόχους, δηλαδή ορισμός των διαφόρων ε, παραπτωμάτων, αδικημάτων και εγκλημάτων, συγκεκριμένες ποινές και άρα ενισχυμένη προστασία των θυμάτων. Παιδική πορνογραφία. Σε αυτή τη φάση τόσο η οδηγία όσο και τη σύμβαση συμφωνούν για τον ορισμό της του παιδιού. Είναι ε, κάτω των 18 ετών. Και αυτό θα πρέπει να είναι συνεπές ολόκληρο το σχέδιο οδηγία, ωστόσο προχωρά περισσότερο από τη σύμβαση όταν ορίζει η παιδική πορνογραφία. Είναι η σεξουαλική φύση του υλικού που είναι κλειδί δεν ορίζεται η σεξουαλική η φύση, η φύση της εκμετάλλευσης του περιεχομένου. δεν υπάρχει διάκριση αυτή τη στιγμή ανάμεσα σε πραγματικές και μη πραγματικές εικόνες ε, κακοποίησης ή εκμετάλλευσης παιδιού. Ωστόσο, ίσως η πιο βασική διαφορά ανάμεσα στα δύο αυτά μέσα είναι η κίνηση στο άρθρο 21 που προβλέπει άμεση δράση από τα κράτη-μέλη ώστε να ε, προχωρήσουν σε μπλοκάρισμα ή σε φιλτράρισμα ώστε να απαγορεύσουν πρόσβαση στην επικράτειά τους σε site τα οποία έχουν παιδική πορνογραφία πολύ ευρεία διάταξη, προχωρά πολύ περισσότερο από τη σύμβαση αλλά δεν δίνει οδηγίες για το πώς προβλέπεται να γίνει η εφαρμογή της. Ίσως αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε περισσότερο. Το μπλοκάρισμα του ίντερνετ δεν συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της σύμβασης ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης για την παρεμπόδιση της σεξουαλικής ε, εκμετάλλευσης των παιδιών, γιατί κανένας από τους ε, συμμετέχοντες δεν το ανέφερε. Ωστόσο, παραπέμπουμε στις νομικές και δημοκρατικές επιπτώσεις μιας τέτοιας ενέργειας. Και θα ήθελα να θυμίσω ότι η εφαρμογή τέτοιων μέτρων θα πρέπει να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα που είναι εγγυημένα στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ιδιαίτερα το δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, την ελευθερία έκφρασης, αλλά επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως τα δικαιώματα των παιδιών προστατεύονται. Το μπλοκάρισμα της πρόσβασης ε, καλεί διεθνή διεθνή ανταπόκριση και το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, αποτελεί το νομικό πλαίσιο για την διεθνή καταπολέμηση. Θα μπορούσαμε λοιπόν να παρέχουμε τη βάση για να εξετάσουμε μορφές μπλοκαρίσματος, τρόπους μπλοκαρίσματος και να καλέσουμε σε διεθνή συνεργασία. Πριν από την ακρόαση μου ζητήθηκε να αναφέρω επίσης τη διάταξη της δικής μας σύμβασης για τη δικαιοδοσία. Τα μέρη θα πρέπει να εισάγουν στις εθνικές τους νομικές διατάξεις τις, ε, τις δυνατότητες ποινική δίωξης. Εκεί αναφέρονται τα θέματα της επικράτειας, της εδαφικότητας, ε, παραπτώματα τα οποία έχουν γίνει σε πλοία ή σε αεροσκάφη, τα οποία είναι γεγραμμένα, ε, νιολογημένα στο εν λόγω κράτος και εκτός από την περίπτωση του κανόνα της εδαφικότητας υπάρχουν κάποιες φορές δυνατότητες επιφύλαξης. Η σύμβαση προβλέπει διάφορα κριτήρια καθώς και απαιτεί ο δράστης και το θύμα να έχουν την ε, κατοικία τους στην επικράτεια του εν λόγω κράτους αν και αυτές οι διατάξεις είναι προαιρετικές και μπορούν να αποτελέσουν και αντικείμενο επιφύλαξης είναι ένα πολύ θαραλέο βήμα και για να μπορούμε να καταπολεμήσουμε και το σεξουαλικό τουρισμό προβλέπουμε την άρση των συνηθισμένων εμποδίων για σεβαρές σεξουαλικά ε, κλίματα που γίνονται στο εξωτερικό και λόγω της εξαιρετικής του η μπορεί αυτό να αποτελέσει αντικείμενο επιφύλαξη και να περιορίσει έτσι το πεδίο εφαρμογή σε σεξουαλικέ ε, ε, πράξεις. Ε, τώρα, όσον αφορά την προστασία του θύματο, είναι πολύ σημαντικό η οδηγία να μιλήσει για δομέ, φιλικές προς τα παιδιά, ώστε να βοηθηθούν τα παιδιά θύματα από τη στιγμή που έχει υπάρξει βία η σεξουαλική παρενόχληση. Είναι πολύ σημαντικό να ληφθεί υπόψη η άποψη ότι οι απόψεις των παιδιών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι επίσης. Um, και έτσι τώρα έρχομαι στην ε, προηγούμενη πρόσκληση της κυρίας Αντζελίλη. Εμείς θέλουμε να δώσουμε και να συμβάλλουμε στην, ε, στο σχέδιο που Θα σας δώσουμε ένα πλήρες κείμενο το οποίο θα συγκρίνει τη σύμβαση και το σχέδιο της οδηγίας. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε αυτό να σας το δώσουμε στις επόμενες εβδομάδες ε, και έτσι φτάνω στο μέλλον και στις, ε, στην επερχόμενη εκστρατεία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ελπίζω ότι αυτό θα σας ε, παρακινήσει ώστε να περάσει η οδηγία από τις διάφορες επικίνδυνες στροφές που έχετε μπροστά σας και αυτό με κάποιο θάρρος. Στις 29 Νοεμβρίου το Συμβούλιο θα ξεκινήσει την εκστρατεία για το σταμάτημα της σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών στη Ρώμη στην Ιταλία. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να δρούμε, να ενημερώνουμε και να φροντίζουμε έτσι ώστε θα δημιουργούνται οι κατάλληλε προποθέσει ώστε να παρεμποδιστούν αυτά τα τρομακτικά γεγονότα που σα ανέφερα πριν, ότι ένα στα πέντε παιδιά είναι θύματα σεξουαλική παρενόκληση και το 80% από αυτά μέσα στον κύκλο εμπιστοσύνη του. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αρχίσουν να επικυρώνουν την σύμβαση ε, και θα πρέπει να πιέσουμε στο αυτό να γίνει γρήγορα, να γίνει εκστρατεία σε εθνικό επίπεδο. Θα ωφεληθούμε από το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, και το, ε, τα τον εστιασμό στα δικαιώματα του παιδιού. Έχουμε βοήθεια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ΜΚΟ, τον Ombudsman, γενική κινητοποίηση σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να γίνει. Θα βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να οργανωθούν, να φτιάξουν τις εκστρατείες, να επικυρώσουν όμως και τη σύμβαση και να αρχίσουν και να τις εφαρμόζουν αυτές. Τα παιδιά είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής της εκστρατείας και η συμμετοχή στην εκστρατεία είναι πολύ σημαντική. Σύμφωνα με τη σύμβαση και το τελευταίο σχόλιο για το άρθρο 12. Στόχος είναι να συνειδητοποιήσει το ευρύ κοινό οι γονείς την ύπαρξη αυτής της βίας και να σπάσουν τα ταμπού, να σπάσει η σιωπή γύρω από αυτού του είδους τα εγκλήματα. Καθημερινά έχουμε νέα νέων θυμάτων σεξουαλικής βίας. Αυτό μπορεί να σας κάνει να σκεφτείτε ότι όλοι γνωρίζουν πως συμβαίνουν όλα αυτά. Ίσως, αλλά εμεί πιστεύουμε ότι πρέπει να εξηγήσουμε τον κίνδυνο αυτό στα παιδιά μας, να τους βοηθήσουμε, να τους μάθουμε να σπάσουν τη σιωπή και να ε, πούν ότι του συμβαίνει. Οι γονείς θα πρέπει να παίξουν δραστήριο ρόλο σε αυτή την ε, ενημέρωση και εκτίμησε αυτό που είπε κάποιος προηγουμένως ότι πρέπει να μιλήσουμε για σεξουαλική αγωγή. Για τους περισσότερους γονείς, οι περισσότεροι γονείς θέλουν να προστατέψουν τα παιδιά τους και δεν θέλουν να μιλήσουν για την σεξουαλικότητα σε πρώιμο στάδιο, σε μικρή ηλικία. Αλλά πρέπει να βοηθήσουμε εμείς τους γονείς να μιλήσουν και εκείνοι με τη σειρά τους για όλα αυτά στα παιδιά τους. Γι' αυτό το λόγο εμείς στο Συμβούλιο της Ευρώπης αναπτύσσουμε ένα πολύ ωραίο εργαλείο child focus για τους γονείς και τα παιδιά που θα τους βοηθήσουν να μιλήσουν. Αυτή η εκστρατεία μπορεί να προκαλέσει δημόσια συζήτηση σε κάποιες χώρες. Θα χρειαστεί να έχουν όλοι θάρρος και εγώ βασίζομαι σε εσά ως ευρωβουλευτές να ηγηθείτε να δώσετε αυτό το θάρρος στους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων, στους εκπαιδευτές, στους γονείς και στα παιδιά. Γιατί δεν θέλουμε αυτή η εκστρατεία να μείνει μυστική. Thank you very much. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα... Ο λόγος για μια σύντομη συζήτηση, σας παρακαλώ γιατί έχουμε καθυστερήσει λίγο, καταρχάς στην κυρία Ζίπελ και μετά στην κυρία Μποσκούρτ. Κυρία Ζίπελ. Ευχαριστώ. Όσο περισσότερο ακούω τους εμπειρογνώμονες, δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ο στόχος της οδηγίας. Άκουσα τον εκπρόσωπο της Eurojust και αναρωτιέμαι πού είναι δηλαδή η προστιθέμενη αξία αυτής της οδηγίας. Σε ποιο ακριβώ σημείο παρεμβαίνει η, η οδηγία. Θέλουμε δηλαδή να καλύψουμε το, το κενό του τι γίνεται στο ίντερνετ με την οδηγία αυτή. Επίσης, θα ήθελα αυτά τα στατιστικά που είπατε, πόσα, ε, πόσες ε, κολάσιμες πράξεις υπάρχουν, πόσα εγκλήματα υπάρχουν. Είπατε πόσα, πόσες εικόνες υπάρχουν, πόσες φωτογραφίες υπάρχουν στο ίντερνετ. Ωραία, αλλά ως τάξη μεγέθους τι παίρνουμε. Δηλαδή μιλούμε για αύξηση των... Ε, των εγκλημάτων ή απλώς αντιγράφονται οι εικόνες και απλώς πολλαπλασιάζονται. Δηλαδή, πού είναι η σχέση, ο συσχετισμός εδώ. Δεν ήταν σαφές. Και η Europol και η Eurojust θα ήθελα να μου πούνε ξεκάθαρα το τι γίνεται με τις ποινικέ απαιτήσει για τα νομικά πρόσωπα. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολος ο τομέας αυτός. Και επίσης, για την πρόληψη σε ό,τι αφορά την ε, σεξουαλική αυτοδιάθεση. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, αλλά δεν νομίζω ότι πάμε όσο μακριά πρέπει. Τα παιδιά που είναι, ε, τα παιδιά που πλήττονται είναι περισσότερο τα παιδιά που έρχονται από ένα ε, ασφαλές περιβάλλον, από ένα κοινωνικό περίγυρο και δεν, δεν μπορούν να πούνε όχι, δεν ξέρουν να πούνε όχι. Κάποιος ε, περνάει στο δρόμο, τους, ε, τους δίνει μια καραμέλα, τους λέει έλα μαζί μου. Ε, αυτό εκεί πρέπει να παρέμβουμε εμείς, να, να μάθουμε το παιδί να λέει όχι. Καλές είναι και οι αλλά νομίζω ότι θα ήταν καλό αν μπορούσαμε να είχαμε χρόνο για να δούμε ποια είναι αντικειμενικά η προστιθέμενη αξία για τη μείωση των εγκλημάτων κατά παιδιών με βάση αυτή την οδηγία. Γιατί σήμερα πραγματικά δεν το κατάλαβα. Ευχαριστώ. Κύριε Μποσκούρτ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω κι εγώ κάποιες ερωτήσεις ε, για τον εκπρόσωπο της Eurojust και για τον εκπρόσωπο της Europol. Καταρχάς, η επιτήρηση και εντοπισμός των παιδιών Μέχρι τώρα μιλάμε για παιδιά τα οποία πέφτουν παγίδα, που είναι θύματα, ε, θύματα εκβιασμού. Πώς ρυθμίζονται στην οδηγία αυτή ε, το θέμα αυτό. Πρέπει να βοηθήσουμε τα ανήλικα παιδιά ώστε να μην πέσουν θύματα αυτών των φαινομένων. Κάπου χάνω τους συνδέσμους. Επίσης θα πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται με τα θέματα των προθεσμιών και με το πότε ακριβώς καταδικάζεται ένα δίκημα και ένα έγκλημα. Ε, και να στραφώ τώρα στον εκπρόσωπο της Eurojust. Ε, σκέφτομαι ε, τα θέματα των κληρικών, την Καθολική Εκκλησία, τις αποκαλέψεις που είχαμε στον τομέα αυτό για τις κακοποίησεις παιδιών. Τι κάνετε σε σχέση με αυτά τα οποία συνέβησαν στην Ιρλανδία, όπου το θέμα απλώς αποσιοποιήθηκε και ο ένας ιερέας απλώς μεταφέρθηκε στη Γερμανία. Νομίζω ότι η Eurojust μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο εδώ. Εσείς τι πιστεύετε, πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει κάτι. Ε, και Πιστεύετε ότι υπάρχει σαφήνεια σε θέματα ε, διαμεθοριακής ε, προστασίας των παιδιών. Υπάρχει δυνατότητα να γίνει κάτι και αν όχι γιατί δεν μπορεί να γίνει και αν ε, ναι τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ευχαριστώ κύριε Μποσκούρτ. Μήπως θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με τον κύριο Λορέλ. Θα απαντήσω καταρχάς στην ερώτηση για το επιπρόσθετο όφελος που έχει να δώσει Eurojust. Η Eurojust δεν ασχολείται με όλα όσα βρίσκονται στην οδηγία. Εμείς είμαστε ένας οργανισμός που συντονίζει δράσεις μεταξύ των χωρών. Δεν ελαμβάνουμε ίδια πρωτοβουλία. Αυτό σημαίνει ότι θα μας ε, ε, εντοπίσει ένας εξαγγελέας από μία χώρα ή εισαγγελεί από χώρες μέλη που εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση και εμείς θα δράσουμε κατόπιν ετήματος από το κράτος μέλος ή από μία αρχή του κράτους μέλους. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα προσφύγουμε εμείς στο δικαστήριο. Αν θέλετε είμαστε ο σύνδεσμος μεταξύ κράτους μέλους και αρχών ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμεί είναι τα θέματα δικαιοδοσίας. Γι' αυτό ακριβώς ε, επεσήμενα και πόσο σημαντικό είναι το θέμα της εξαοεδαφικότητας και της εξοεδαφικής ε, δικαιοδοσίας. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι μπορούμε εμείς ή οι εισαγγελίε στα κράτη-μέλη μπορούν να ε, διώξουν για ένα έγκλημα το οποίο έχει διαπραχθεί εκτός της χώρας στην οποία βρίσκεται ο δράστης. όλα όσα περιγράφονται στην οδηγία δεν αφορούν τις δικές μας εργασίες. Εμείς μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και χωρίς αυτή την οδηγία, αλλά σαφώς θα υπάρχουν ε, επιπτώσεις για τους εισαγγελείς που ασχολούνται με τα ε, αδικήματα αυτά στα κράτη-μέλη. Υπήρχε μια ερώτηση για τον αριθμό των φωτογραφιών και τον αριθμό των θυμάτων. Υπάρχουν πάρα πολλά θύματα στην υπόθεση που σας ανέφερα. Σε μία χώρα είχαμε 7 θύματα, αλλά υπάρχουν και πολλά θύματα σε όλες τις χώρες που ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Οι φωτογραφίες όμως δεν είναι όλες φωτογραφίες των θυμάτων που εντοπίστηκαν και που κακοποιήθηκαν από τους δράστες αυτής της υπόθεσης. Όπως αναφέρθηκε ε, σήμερα το απόγευμα, θα αναρτώνται φωτογραφίες στο διαδίκτυο και θα κυκλοφορούν συνεχώς και πολλές από αυτές τις φωτογραφίες ε, είναι γνωστές εκ των προτέρων. Το δίκτυο όμως που περιέγραψα ε, παρήγαγαν νέες φωτογραφίες. είχαμε συλλήψεις και κατασχέσεις στα κράτη-μέλη και στις κατασχέσεις ε, μεταξύ των φωτογραφιών που βρέθηκαν είχαμε φωτογραφίες και πολλών άλλων παιδιών πέραν των θυμάτων που εντοπίσαμε εμείς. Τώρα, για την πολυμερή συνεργασία, τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. από πλευρά μα δεν θα έχουμε σοβαρέ συνέπειε με, λόγω τη οδηγία. Όπως σα είπα και πριν, θα είναι κάτι το οποίο θα έχει ε, περισσότερο επίπτωση στις έρευνε, στα κράτη-μέλη. Αν για παράδειγμα δεν υπάρχει ανάγκη ε, κατηγορίας εκ μέρου του θύματο που σημαίνει ότι μία αρχή σε ένα κράτο μέλος μπορεί να ξεκινήσει έρευνα χωρίς να προσφύγει κάποιο στις αρχές, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε για παράδειγμα την έναρξη μιας επιχείρησης μεγάλης κλίμακας την οποία θα συντονίσει η Eurojust. Όλα κατά κάποιο τρόπο είναι αλληλένδετα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Σέρτη. Ευχαριστώ πολύ και εγώ και θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά που μόλις είπε ο συνάδελφος από τη Eurojust. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες φωτογραφίες παιδιών τα οποία αποτελούν αντικείμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Κάποιες είναι παλιές φωτογραφίες, κάποιες είναι καινούριε. Και όταν ε, ε, βάζουμε σε κλίμακα του εγκληματίε, έχουμε το κατώτερο σκαλοπάτι και έχουμε και το ανώτερο. Κάποιοι από αυτού του ανθρώπους απλώς απολαμβάνουν να τις ε, κοιτούν. Ε, κάποιοι τις παράγουν, κάποιοι έχουν στούντιο με ε, κάμερες οι οποίες ε, ε, λειτουργούν σε ζωντανή μετάδοση και μπορεί να ζητήσει κάποιο από το παιδί να κάνει κάτι και εσύ να το απολαύσει από την άλλη άκρη τη οθόνη. Ή επίσης μπορεί ε, να υπάρχει και διαβατήριο για να μπει σε, σε συζήτηση, σε chat rooms τα οποία είναι μυστικά, αλλά σε κάποιες άλλες περιπτώσεις δεν χρειάζεται καν password, είσαι απλά ως μέλος της ομάδας και ε, εκτός από τις παλιές φωτογραφίες υπάρχουν και νέες φωτογραφίες. Εδώ αναφερόμαστε σε βιασμό παιδιών και ουσιαστικά το ίντερνετ κάνει διευκόλυνση αυτής της διαδικασία. Τα βασικά, αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι οι βιασμοί των παιδιών. Το διαδίκτυο ε, διευκολύνει τους δράστες και τους κρύβει κιόλα. και επίσης τους επιτρέπει ε, να ε, διαδίδουν αυτά τα, τα στοιχεία και με εκπλήσει το γεγονός ότι κάθε χρόνο παρά το γεγονός ότι γνωρίζουν ότι έχουμε μέσα στο διαδίκτυο ε, συλλαμβάνονται ε, δάσκαλοι, ιερείς, ε, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε συλλαμβάνουμε. Όσον αφορά την οδηγία, τίποτα δεν είναι τέλειο, αλλά είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, διότι βοηθά τα κράτη-μέλη να συντονίσουν τις προσπάθειές τους και να μπορέσουμε να κάνουμε μια επιπλέον προσπάθεια για τις συνδυασμένε δράσεις μας. Και πρέπει φυσικά να γίνει ένα βήμα περαιτέρα και ένα ακόμα βήμα με βάση το αρχικό στάδιο αυτό. Αλλά νομίζω ότι θα βοηθήσει και εμά και τα κράτη-μέλη αυτή η οδηγία. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Madam. Ευχαριστώ. Ένα από τα ερωτήματα ήταν η προστιθέμενη αξία για τα πρότυπα και τους μηχανισμούς που έχουμε μέσω αυτής της οδηγίας. Ίσως ε, να μην ήταν ε, προς εμένα η ε, ερώτηση, αλλά θα επιχείσω και εγώ αυτά που είπε ο κύριος που κάθεται δίπλα μου, γιατί νομίζω ότι όντως αυτό το θέμα είναι θέμα συνεργασίας. Έχουμε τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, που είναι μια εξαιρετική βάση για να δουλέψουμε. Έχουμε την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οδηγιών που θα είναι άμεσα εφαρμόσιμες αλλά θα ήθελα να ε, σας βεβαιώσω ότι το σχέδιο οδηγίας θα προχωρήσει πέρα από τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης και δεν θα επηρεάσει το πεδίο εφαρμογής, ούτε θα το περιορίσει τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης το οποίο θα μπορούσε να μπλοκάρει την ε, υπογραφή από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβουλίο της Ευρώπης αποτελείται από 47 κράτη-μέλη. Αυτό μας δίνει την ευκαιρία να συνεργαστούμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε, είναι σημαντικό νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση από κοινού με άλλους διεθνείς οργανισμούς να συνεργαστεί και ελπίζω με την οδηγία αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση να το πράξει και να υπάρξει προστιθέμενη αξία γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Ευχαριστώ. Okay. Thank you. Uh, Εγώ ευχαριστώ. Τώρα, θέλω ότι πρέπει να προχωρήσουμε στο τρίτο πάνελ και ζητώ τους ομιλητές, την κυρία Μπανώτη, Η κυρία Μπάρν και την κυρία Μάλα να έρθουν εδώ στο Προεδρείο να καθίσουν. Ας ξεκινήσουμε το τρίτο μέρος που σχετίζεται με τις διεθνείς προοπτικές. Ξεκινώντας με την κυρία Μαάλα, που είναι η συγγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για το θέμα της παιδικής πορνογραφίας και της παιδικής πορνείας. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Έχω την τιμή να απευθύνομαι σε εσά σε αυτή τη συνεδρίαση που είναι αφιερωμένη στην οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που στόχο έχει την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης ε, των παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας. Ε, ε, λόγω της φύσης της εντολής μου, κάθε σκέψη, δράση που στοχεύει στην πρόληψη και στην καταπολέμηση αυτών των φαινομένων με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρον. Το Σεπτέμβριο 2009, κατά τη διάρκεια της 12ης Συνόδου του Συμβουλίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, παρουσίασα μια έκθεση για την πορνογραφία την παιδική και τον Οκτώβριο του 2010 θα παρουσιάσω στη Γενική Συνέλευση της Νέας Υόρκης μια έκθεση για την εξέλιξη της υιοθεσία και της εφαρμογής του προαιρετικού πρωτοκόλλου για την πώληση παιδιών, την, πορνεία, την εκπόρνευση παιδιών και την πορνογραφία παιδιών που σας θυμίζω ε, ε, ε, ολοκληρώνει μία δεκαετία επιτρέψατε μου να μοιραστώ μαζί σας κάποιες απιστώσεις σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Το φαινόμενο αυτό που θεωρείται έγκλημα, μία από τις χειρότερες μορφές παραβίασης του δικαιώματος, των δικαιωμάτων των παιδιών και μεγάλη ε, προσβολή στην ακυριότητα και στην αξιοπρέπεια των παιδιών, πολλοί μηχανισμοί και μέσα έχουν ε, θεσπιστεί με πρώτη και καλύτερη την ε, Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών. Το πρωτόκολλο είναι προαιρετικό για την πώληση, την πορνεία και την πορνογραφία και ένα σωρό άλλα μέσα όπου συμμετέχουν διάφορα χώρες χωρίς να ξεχνάμε την πρόσφατη δήλωση και έκκληση σε δράση του Ρίου του περασμένο Νοέμβριο. Όλα σε αυτές τις δεσμεύσεις έχουν επιτρέψει να σημειωθούν σημαντικές πρόοδοι. Πολλές πρωτοβουλίες σε ιδιωτικό, δημόσιο τομέα, μικείο, ε, οργανισμοί που συχνά συνεργάζονται σε διεθνές επίπεδο, σε περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο για να προλάβουν και να καταπολεμήσουν το φαινόμενο αυτό, έχουν οδηγήσει στην ε, μείωση του φαινομένου. Ωστόσο, ε, έχουμε πολλές προκλήσεις όσον αφορά τη γνώση της πραγματικότητας ταυτότητας στο φαινόμενο, την πρόληψη και την, προ... την πρόληψη του φαινομένου. Ένα, μια πρώτη πρόκληση είναι σχετική με το εύρος και τις ε, εξελικτικές τάσεις. Πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία που λαμβάνουμε, φαίνεται σαφώς πως ορισμένες μορφές, όπως ο σεξουαλικός τουρισμός, η πορνεία παιδιών, η παιδοπορνογραφία μέσω του ίντερνετ, οι τηλεπικοινωνίες, οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις μέσω κοινωνικών δικτύων αυξάνονται σε σημαντικό βαθμό και πολλά παιδιά, κορίτσια και αγόρια παραμένουν θύματα τέτοιων μορφών σεξουαλικής εκμετάλλευσης ολόκληρο τον κόσμο. Οι εικόνες σεξουαλικά ε, ε, κακοποιημένων παιδιών είναι όλο και πιο σοκαριστικές και βίες και τα παιδιά στις φωτογραφίες είναι όλο και πιο μικρά. Είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε πόσε εικόνε κυκλοφορούν λόγω τη διαθεσιμότητα αυτού του παιδοπορνογραφικού υλικού σε κοινωνικά δίκτυα ε, και σε δίκτυα παιδοφιλίας. Ε, βλέπουμε επίσης πολύ συχνά να καλούνται, να παρελοχνούνται τα παιδιά στο ίντερνετ μέσω του grooming όπως αποκαλείται. Ωστόσο είναι δύσκολο ακόμα να καθορίσουμε ε, την ακριβή φύση. Είναι δύσκολο να εντοπίσουμε τα παιδιά θύματα. Είναι διεθνής η διάσταση του φαινομένου. Δεν αρκεί δεν είναι επαρκή ο συντονισμό ανάμεσα στου διάφορου φορείς όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών είναι επίσης μικρός ο αριθμός των περιπτώσεων που αναφέρονται ε, από τα θύματα ή από, ε, από τις οικογένειές τους. Συχνά λόγω ατελών νομοθεσιών και μη, μη συστηματικής προσφυγής στη δικαιοσύνη, δυσκολία ανά της πρόγραμβασης στην δικαιοσύνη, στους μηχανισμούς προσφυγής και πολλές φορές ε, λόγος της μη αναφοράς είναι το κόστος της δικαστικής διαδικασίας. Και πάλι ενώ όλοι, όλοι συμφωνούν στο ότι είναι πολύ περίπλοκο αυτό το φαινόμενο με, λόγω του ότι έχει πολλαπλές μορφές και πολλούς παράγοντες που συχνά αλληλοσυνδέονται και που επιδεινώνουν την, ε, την ε, τροτό χαρακτήρα των παιδιών. Η φτώχεια, οι κοινωνικές ανισότητες, οι ορισμένες κοινωνικοί κανόνες, ε, υποβάθμιση του περιβάλλοντος το AIDS, μετακίνηση πληθυσμών, οι ένοπλες συγκρούσεις και άλλες επίγουσες καταστάσεις, η άνετη πρόσβαση στις τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας και φυσικά μια κλιματικότητα όλο ένα και πιο οργανωμένη, αλλά και μια ετατική ζήτηση, μια μόνιμη και στεναρή ζήτηση της, που, που υποστηρίζεται από τη βιομηχανία της, του σεξ. Και τέλος, βλέπουμε πολύ και διαπιστώνουμε τον αυξανόμενο αριθμό κατηγοριών παιδιών που είναι πολύ ευάλωτα, όπως ε, τα μη συνοδευόμενα παιδιά που μεταναστεύουν, τα παιδιά των δρόμων, τα παιδιά που υιοθετούνται παράνομα, τα παιδιά που είναι θύματα πώληση ή εμπορίας, τα ε, παιδιά που εργάζονται, τα ανάπηρα παιδιά ή τα παιδιά που είναι σε ιδρύματα ή σε σοφρονιστήρια, τα παιδιά που έχουν διάφορες, ε, διάφορους εθισμούς όπως ναρκωτικά ή αλκοόλ. Το πολύ σημαντικό θέμα είναι οι συνέπειε για αυτά τα παιδιά, που είναι σωματική, ψυχική και κοινωνική φύση, μεταδοτικέ ασθένειε, AIDS, πρώιμε ε, εγκυμοσύνε. Ε, ε, συμπεριφορές εθιστικές, στιγματισμός κοινωνικός και περιθωριοποίηση. Κάτι ακόμα που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε είναι η διάδοση των εικόνων περδοπορνογραφίας μέσω του ίντερνετ και των τηλεπικοινωνιών που επιπλέκουν ε, τις ε, συνέπειες ε, των καταχρήσεων προς τα παιδιά και επιφέρουν αντίκτυπο στην αποκατάσταση των θυμάτων. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα εικόνα των παιδιών και των κακοποιημένων δεν θα εξαφανιστούν ποτέ από το ίντερνετ, πράγμα που έχει καταστροφικές επιπτώσεις για τα θύματα. Κάτι άλλο που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι τα παιδιά μπορεί να πέσουν θύματα πορνογραφίας, αλλά εκτίθενται επίσης και η έκθεση των παιδιών στην παιδοπορνογραφία επηρεάζει και εμπνέει τις σεξουαλικές πρακτικές των νέων. Και οι, πορνογρα... και οι πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η πορνογραφία πολύ συχνά είναι ο βασικός χώρος ε, σεξουαλικής αγωγής για τους νέους. Διευκολύνει αυτό τη γενίκευση συμπεριφορών που συνδέονται με την πορνογραφία. Όσον αφορά τις απαντήσεις των κρατών για τα θέματα πρόληψης και προστασίας αυτών των παιδιών, εναντίον αυτών των, των ε, πρακτικών, όσον αφορά τις επικυρώσεις, είναι χωρίς αμφιβολία αυξάνονται οι επικυρώσεις ε, για τους ε, διεθνείς και περιφερειακούς μηχανισμούς. Θα σας θυμίσω ότι μέχρι στιγμής 137 κράτη εταίροι έχουν επικυρώσει το προαιρετικό πρωτόκολλο που σχετίζεται με την πώληση, την παιδιών, την παιδική πορνεία και πορνογραφία. 22 χώρες της Ένωσης έχουν υπογράψει το πρωτόκολλο, αλλά 4 χώρες δεν έχουν ακόμα επικυρώσει, ενώ το έχουν υπογράψει. Τσεχία, Ιρλανδία και Μάλτα. Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία από την εκμετάλλευση και τις σεξουαλικές καταχρήσεις που άρχισε να ισχύει το 2010, μόνο 8 χώρες την έχουν επικυρώσει, από τις οποίες οι πέντε είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι συμβαίνει. Εντάξει, καλό είναι να υπογράφει και να επικυρώνει τι συμβάσει, αλλά καλύτερο είναι όταν υπάρχει μια πραγματική επιβολή τη νομοθεσία. Διαπιστώνουμε σε όλε τι χώρε ότι έχουν γίνει πολλέ νομοθετικέ μεταρρυθμίσει. Ωστόσο, παρά τι προσπάθειε, πολλά πρέπει να γίνουν. Γιατί υπάρχουν πολλέ νομικέ ανεπάρκειε. Ορισμένε εθνικέ νομοθεσίε ε, υπάρχουν, αλλά ορισμένε δεν ορίζουν ακριβώ τι παραβάσει και δεν ποινικοποιούν, δεν τιμωρούν όλε τι μορφέ εκμετάλλευση ορισμένες άλλες τιμωρούν, ή ποινικοποιούν τις, τη σεξουαλική κακοποίηση. Άλλοι δεν προβλέπουν την ιατροδικαστική βοήθεια για τα παιδιά. Δεν θεσπίζουν έξω εδαφικές αρμοδιότητες όσον αφορά την ε, σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών. Και όσον αφορά την νομοθεσία πάντοτε, πολλές χώρες δεν διαθέτουν αποτελεσματικό και εύκολα προσβάσιμο σύστημα, γιατί πρέπει να μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ώστε να επιτρέπουν την ενημέρωση ε, για την σεξουαλική παρενόχληση και την παρακολούθηση αυτών των παιδιών. Αυτό σημαίνει, βέβαια ότι και οι παραβάτες αλλάζουν χώρα κάθε φορά που ζορίζουν τα πράγματα και πάνε εκεί που είναι πιο ήπια η νομοθεσία, πιο επίκης. Τώρα, πολλά προγράμματα δράσης, στρατηγικές ε, και υπηρεσίες έχουν δημιουργηθεί αλλά δεν αρκούν. Συχνά είναι περιορισμένα γεωγραφικά ή χρονικά όλα αυτά. Σε θέματα πρόληψης, πολλές εκστρατείες ευαισθητοποίησης και εργαλεία ενημέρωσης έχουν γίνει. Δυστυχώς, συχνά είναι εξτρατείες ε, συγκυριακές και δεν μετράται ο αντίκτυπός τους. Όσον αφορά την πρόσβαση στα πορνο, πορνογραφικά site, ε, έχουν διεφτιαχτεί μηχανισμοί ελέγχου, safer internet και διάφορα άλλα για να προληφθεί ο σεξουαλικός τουρισμός έχει υπάρξει και έλεγχο των τουριστικών site ωστόσο όλα αυτά είναι περιορισμένα σε ορισμένες χώρες και συχνά είναι οι πιο ε, προηγμένες βιομηχανικά χώρες. Παρά την μεγαλύτερη ερωτότητα των παιδιών, έχουμε το Youth Advisory Council, το Peer-to-Peer Education, αλλά πρέπει ακόμα να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την πρόσβαση των παιδιών στην ενημέρωση, την την ε, φροντίδα των παιδιών θυμάτων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και την λήψη υπόψη των αναπόψεων των παιδιών κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των διαδικασιών. Γιατί σας το θυμίζω ότι τα παιδιά θεωρούνται νέα οστήματα αλλά κυρίως ως φορείς και αποτελούν τμήμα αναπόσπαστο της λύσης. Τώρα, όσον αφορά την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, πολλέ από αυτέ έχουν υιοθετήσει κώδικε διοντολογία, έχουν ξεκινήσει εκστρατείε, προγράμματα ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Κράτη έχουν ε, υιοθετήσει νομοθεσίε που ε, αναθέτουν ε, την ευθύνη στου σερβερ, στι τραπεζικέ επίση επιχειρήσει Αλλά αυτό θα πρέπει να επηρεάσει όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις μεταφορών και ούτω καθεξής. Τώρα, υπάρχουν, ε, υπάρχει διεθνή συνεργασία, διευκολύνεται η συνεργασία των ε, αστυνομικών δυνάμεων, έχουν αναφερθεί παδείγματα η Virtual Global Task Force, Internal Watch Foundation, η Europol, η ε, Eurojust κτλ. Αλλά όλοι αυτοί οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες διευκολύνουν το συντονισμό σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, αλλά πολύ καλό θα ήταν να ενισχυθούν και να γενικευθούν γιατί το φαινόμενο της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ξεπερνά τα σύνορα. Ένα, μια τελική διαπίστωση τι συμβαίνει με την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση. Σα θυμίζω ότι όλοι όσοι έχουν υπογράψει την Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού έχουν ε, δεσμευτεί για να έχουν μηχανισμού παρακολούθηση και προστασία των παιδιών. Ωστόσο, πολλέ χώρε δεν έχουν ακόμα αυτό το μηχανισμό και είναι πάρα πολύ δύσκολο να μετρήσουμε τι εξελίξει. Μετά από όλες αυτές τις γενικές διαπιστώσεις επιτρέψατε μου να μιλήσω για την οδηγία. Εν γέννη αυτή η οδηγία όταν τη διάβασα Εμένα μου φάνηκε πως είναι μια απάντηση στις ε, διαπιστώσεις που σας ανέφερα, γιατί θέλει να ε, συμπληρώσει και να αρμονίσει την νομοθεσία με τα περιφερειακά και διεθνή μέσα, τα οποία είναι ήδη επικυρωμένα, και να προσεγγίζει τις νομοθετικές ε, διατάξεις που ισχύουν στο διάφορα κράτη-μέλη, ενσωματώνοντας και το ποινικό δίκαιο. Σαφείς ε, επίσης ορισμοί περιλαμβάνονται για όλες τις μορφές ε, σεξουαλικής ε, παρενόχλησης και εκμετάλλευσης του παιδιού. Εν γέννη, αυτή η οδηγία ανταποκρίνεται σε αυτές τις διαπιστώσεις γιατί στόχο έχει να διευκολύνει τις έρευνες και την έναρξη ανακρίσεων και διώξεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στοχεύει να προστατεύσει τα θύματα με εγγύηση της ιατροδικαστικής και ψυχολογικής βοήθειας και αρρωγής και παρακολούθηση χωρίς να ξεχνάμε και τα μέτρα αποζημίωσης και έχει στόχο λοιπόν να έχει πρόσβαση και να, δώσει, να τονίσει τους πρώην παραβάτες αλλά και να εμποδίσει την πρόσβαση στην πορνογραφία στο ίντερνετ αλλά και να βελτιώσει τη συνεργασία στον τομέα αυτό όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης δεδομένης της, διεθν... διακρατική διάσταση του φαινομένου. Δεν μπορώ λοιπόν να εκφράσω τη χαρά μου που βλέπω αυτή την οδηγία που απαντά και που λαμβάνει υπόψη το συμφέρον του παιδιού λαμβάνει υπόψη όλες τις μορφές και τις εξελικτικές τάσεις του, του φαινομένου, δηλαδή ε, ε, βασίζεται στην προστασία, στην πρόληψη και στη δίωξη και μιλά κυρίως για συντονισμό. Αλλά να επανέλθω για ορισμένα σημεία που νομίζω ότι είναι σημαντικά και ξεκινώντα από το συμφέρον του παιδιού, το πρώτο θέμα είναι το ηλικία του παιδιού. Και όταν διαβάζουμε την οδηγία και διαβάζουμε και τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει, λέμε για παιδιά και υπήρξαν προτάσει να, να μιλήσουμε για ανήλικες κάτω το 18 και μιλάμε και για την ε, ηλικία σεξουαλικής συγκατάθεση να σας πω ότι είναι σημαντικό να σκεφτούμε ότι κανένα παιδί κάτω το 18 δεν είναι σε θέση να συγκατατεθεί ρητά στο να συμμετέχει στην ε, σεξουαλική του εκμετάλλευση που συμπεριλαμβάνει και πορνογραφικές ε, εικόνες. Αυτή η προσφυγή στην ηλικία του παιδιού έχει νόημα παρά μόνο αν δεν πρόκειται για σεξουαλική εκμετάλλευση. Τώρα, όσον αφορά ένα σημαντικό σημείο, δηλαδή τις δραστηριότητες ανάμεσα στους συνομιλίκους και αναφέρομαι στις διατάξεις του άρθρου 20 της Σύμβασης Λανζαρότη που θα μπορούσε να χρησιμεύσει γιατί κάθε μέρος μπορεί να επιφυλαχθεί του δικαιώματος να μην εφαρμόσει πλήρως ή εν μέρη τις ε, παραβάσεις που σχετίζονται με την παραγωγή και τη διάδοση ε, υλικού που, έχει, ε, που περιλαμβάνει παιδιά με την ηλικία συγκατάθεση, με τη δική του συγκατάθεση και άρα με τη, και μόνο για ιδιωτική χρήση. Άρα εκεί δεν υπάρχει σεξουαλική εκμετάλλευση. Κανένα παιδί που είναι θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευση δεν μπορεί να διωχθεί, ούτε να τιμωρηθεί, ούτε και να κρατηθεί, ούτε και να απελαθεί. Αντιθέτως πρέπει να προστατευτεί και να βοηθηθεί και να αποζημιωθεί σύμφωνα με την αρχή του ε, ανώτερου συμφέροντος του παιδιού. Κάτι ακόμα που είναι σημαντικό είναι οι κυρώσεις, οι ποινές. Είναι επιτακτικής ανάγκης να ξαναδούμε αυτά που υπογραμμίζει η οδηγία, αλλά να ε, είναι πιο, σο, ε, πιο σοβαρές οι ποινές, να είναι αποτρεπτικές και να σας θυμίσω ότι πρόκειται για έγκλημα και σοβαρή παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού να σκληρύνουν οι ποινές με ελάχιστες προδιαγραφές που θα προβλεφθούν και θα επιτρέψουν κάπως να εναρμονιστούν οι απαντήσεις σε ποινικό επίπεδο για όλα τα κράτη-μέλη. Και τέλος να μεριμνήσουμε ότι, ώστε η αρχή της εξοεδαφικότητας να συμπεριληφθεί εδώ. Μια άλλη παρατήρηση και επιμένω εδώ για την προστασία γιατί είναι επιτακτική ανάγκη να έχουμε έναν ωραίο νόμο αλλά να υπάρχουν και πραγματικοί μηχανισμοί προσφυγής να είναι προσβάσιμη όλη αυτή και να επιμείνουμε για την ενίσχυση των διατάξεων και για την προστασία των παιδιών θυμάτων κατά τη διάρκεια των δικαστικών υποθέσεων σεβασμό στις αρχές του συμφέροντος του παιδιού, να ακούγεται το παιδί και να ενημερώνεται για τα δικαιώματά του σε μια γλώσσα που κατανοεί. Και τέλο πάντοτε για την προστασία, η διάσταση αποκατάσταση και παρακολούθησης είναι κεφαλαιόδου σημασία και σα θυμίζω πως οι συνέπειες είναι εξαιρετικά ε, σοβαρές μέσο και πρόθεσμα. Τέλο, όσον αφορά την ε, online πορνογραφία και τη σεξουαλική παρενόκληση online, το grooming, ε, η εξάρθρωση των δικτύων είναι πολύ σημαντική. Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν και να υπάρχει διείσδυση από τις δικαστικές αρχές που έχουν καταρτιστεί κατάλληλα και είναι πρακτικές που ήδη υπάρχουν σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήταν σκόπιμο να επεκταθούν. Τέλος, όσον αφορά το μπλοκάρισμα των site του ίντερνετ και τη διαγραφή των εικόνων, ε, αρκεί, είναι δυσανάλογο, είναι κάτι το εφικτό. Επιτρέψτε μου να μου σας πω είναι εκμετάλλευση, είναι έγκλημα και είναι σοβαρή παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού τα, οι μηχανές ε, έρευνας, ε, οι, οι φορείς της τηλεπικοινωνίας, οι σερβερ θα πρέπει άμεσα να εντοπίζουν το site, να το μπλοκάρουν οι ίδιοι σύμφωνα με κανόνες που θα αριθμιστούν ε, συγκεκριμένα για τους στόχους της δικαστικής έρευνας. Άρα λοιπόν το business θα πρέπει να είναι αυτό το οποίο θα ενημερώσει και να ε, εμποδίσει την πρόσβαση του συγκεκριμένου site και για να διασφαλίσουμε το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή των θυμάτων και να σταματήσουν να κυκλοφορούν οι εικόνες και επιμένω γι' αυτό οι προμηθευτές των υπηρεσιών θα πρέπει να, να, να παρεμποδίζουν την πρόσβαση στα site που, φέρουν αυτές τις, που δείχνουν αυτές τις εικόνες. Έπειτα, οι μηχανισμοί ελέγχου και monitoring και παρακολούθηση έχουν ήδη εφαρμοστεί. Θα πρέπει να διευρυθούν ακόμα περισσότερο και είναι σαφέ πω το μπλοκάρισμα δεν αρκεί δεδομένε της διεθνού διαστάσεως και των εξελίξεων τη τεχνολογία, της ανάπτυξης του οργανωσμένου εγκλήματο, της πρόσβασης ε, της εύκολης ε, ε, της τεχνολογίε τη επικοινωνίας. Όμως είναι κάτι πολύ σημαντικό παρόλα αυτά και να διευκρινίσω και το εξή. Δεν θέλουμε εμείς να τα ρίξουμε όλα στις τεχνολογίες της επικοινωνίας, αλλά να είναι ασφαλισμένη η χρήση των τεχνολογιών αυτών για τα παιδιά και πρέπει να είμαστε αρκετά έξυπνοι να, το χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ίδιες τεχνολογίες για να ενημερώσουμε, να εκπαιδεύσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε, να τονίσουμε, να προειδοποιήσουμε τον κόσμο. Δηλαδή δεν, είναι, το χρησιμοποιούν την επικοινωνία αυτή και τα, το ίντερνετ μόνο αυτά τα αρπακτικά. Σας θυμίζω ότι τα παιδιά είναι αυτά που είναι και τα πιο ε, που είναι το πιθανότερο να ενημερωθούν μέσω των νέων τεχνολογιών γιατί είναι και τα πιο εξοικειωμένα με τις νέες τεχνολογίες. Ανταλλαγή λοιπόν πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε διεθνές επίπεδο γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος για να ανοιχνευτούν οι παραβιάσεις να εντοπιστούν τα παιδιά θύματα και να έχουν αίσιο πέρας οι διώξεις. Και έπειτα το πρόβλημα δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό, είναι διαμεθοριακό, είναι διεθνές και θα πρέπει και στον τομέα της συνεργασίας να μπορούμε να δίνουμε μια βοήθεια και στις χώρες που είναι υπό ανάπτυξη για να μπορέσουν να έχουν τα απαραίτητα συστήματα και τις δεξιότητες. Τέλος, η οδηγία αυτή Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν επαφές ε, τακτικές, θα πρέπει να αναλαμβάνουμε τα παιδιά ή να βλέπουμε τι συμβαίνει με τα παιδιά μετά τα παιδιά θύματα. Να υπάρχει μια κάποια παρακολούθηση. Ε, το ενδιαφέρον αυτή της οδηγίας ξεπερνά το πλαίσιο της απλώς της νομοθεσίας γιατί στοχεύει όπω είπαμε ε, στη δημιουργία ενός συστήματος προστασίας με βάση τη σύμβαση των δικαιωμάτων του παιδιού και κυρίω θέλει να εξασφαλίσει μια αλυσίδα προστασίας όπου οι φορεί συνδέονται μεταξύ τους σε τοπικό, ε, εθνικό και διεθνέ επίπεδο και αποτελεί μια καλή βάση εργασία πρέπει να βελτιωθεί και επιτρέψτε μου κυρία Πρόεδρε να επαναλάβω τις ευχαριστίες μου στους διοργανωτές αυτής της ακρόασης και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω ε, συμβολή ε, που θα μπορούσα να σας προσφέρω. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ε, ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά σας ευχαριστούμε πολύ. Eh, <laughs> για την εξαντλητικότατη παρουσίασή σας. Ελπίζω να μπορέσετε να μου δώσετε και μία διεξοδική έκθεση. Αν έχετε την ευγενή καλοσύνη να τη στείλετε στην γραμματεία, για μας θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι 6 και 10, έχουμε ακόμα δύο παρεμβάσεις και στη συνέχεια θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας ε, στις 6 και μισή το αργότερο Γι' αυτό λοιπόν να δώσω αμέσως το λόγο στη κυρία Μπίρν, η οποία εκπροσωπεί το κέντρο αθών της UNICEF. Uh, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ που καλέσατε τη UNICEF για να παραστεί σε αυτή τη συνεδρίαση. Η UNICEF ε, παγκοσμίως ασχολείται με το θέμα αυτό. Ε, Εγώ προέρχομαι από ένα ερευνητικό κέντρο το οποίο εδρεύει στη Φλωρεντία, στην ε, Ιταλία και Μαζί με τα υπάρχοντα στοιχεία ε, και τις έρευνες που γίνονται έχουμε πολλά στοιχεία για τους ε, παράγοντες κινδύνου. Η πρώτη έρευνα εξετάζει το θέμα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης μέσω του διαδικτύου και άλλων ε, τεχνολογιών επικοινωνίας καθώς επίσης και τα δικήματα κατά παιδιών που διαπράττονται εκτός διαδικτύου αλλά μπορεί να ξεκινήσουν στο διαδίκτυο μέσω grooming και σεξουαλικής παραπλάνησης και το δεύτερο, η δεύτερη έρευνα ασχολείται με τα θέματα θέματα του σεξουαλικού τουρισμού. Καταρχάς να πω το γεγονό ότι τα παιδιά είναι ευάλωτα στα ε, σεξουαλικά αδικήματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις ε, συνθήκες ε, ζωής τους, την ηλικία τους, το οικογενειακό και περιβάλλον τους, αν βρίσκονται σε αστικό υπαίθριο περιβάλλον, την αναπηρία τους και πάρα πολλές άλλες πτυχέ οι οποίε κάνουν τα παιδιά πιο ευάλωτα. Η σεξουαλική κακοποίηση δεν γίνεται μόνο από παιδόφιλους ή ανθρώπους οι οποίοι ε, είναι σεξουαλικά διαστραμμένοι, αλλά άνθρωποι οι οποίοι τους εκμεταλλεύονται ε, στην καθημερινή τους ζωή και εκμεταλλεύονται τις ε, ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες βιώνουν. Ορισμένες φορές άνθρωποι στο στενό οικογενειακό περιβάλλον είναι ε, οι δράστες των σεξουαλικών εγκλημάτων και συνήθω είναι άτομα τα οποία τα παιδιά θεωρούν ότι μπορούν να εμπιστευθούν. Ε, το 80% στι Ηνωμένε Πολιτείε των ε, δραστών είναι άτομα γνωστά στα παιδιά και ένα μεγάλο ποσοστό είναι μέλη τη οικογένεια του και τα στατιστικά στοιχεία είναι αντίστοιχα σε υπόλοιπο, στον υπόλοιπο κόσμο. με την άφηξη του διαδικτύου και των υπόλοιπων τεχνολογιών πληροφορίας έχουν αυξηθεί ε, τα περιστατικά, ε, διότι η αυξημένη πρόσβαση σημαίνει ότι υπάρχει περισσότερη πρόσβαση για τα παιδιά στη γνώση και επικοινωνία με, τους, ε, με άλλα παιδιά της ηλικία τους, αλλά από την άλλη είναι έρμεο τη σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Η κοινωνική μορφή του ίντερνετ δίνει τη δυνατότητα σε πάρα πολλούς ανθρώπους να ε, κάνουν κατάχρηση ε, σε τυχαία βάση. Ο σεξουαλικός τουρισμός επίσης διευκολύνεται λόγω της αύξησης και εξάπλωσης αυτών των νέων τεχνολογιών που διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ε, δραστών που ταξιδεύουν και φυσικά έχει αλλάξει και η αντίληψη που έχουν τα παιδιά μεταξύ των ορίων του εικονικού και του πραγματικού κόσμου διότι για τα παιδιά είναι ή ανύπαρκτα τα όρια ή συγχωνεύονται. Ε, και τα παιδιά είναι πολύ πιο εύκολο να γνωρίσουν άλλου ανθρώπου από ότι οι ενήλικες. Και ο τρόπο με τον οποίο τα παιδιά και οι ενήλικες αντιμετωπίζουν το διαδίκτυο είναι διαφορετικό και αυτό διευρύνει το χάσμα και δυσκολεύει, δυσχεραίνει το ρόλο των ε, γονιών στο πώ να προστατεύσουν τα παιδιά του. Διότι σε ποιον ε, θα στραφούν τα παιδιά όταν έχουν πρόβλημα, με, στους γονείς τους ή στα άλλα παιδιά, στους εικονικούς ή στους πραγματικούς τους φίλους. Βέβαια πολλά παιδιά δεν είναι είναι έρμεα στην εκμετάλλευση, πολλά από αυτά τα παιδιά μπορούν εύκολα να σερφάρουν στο διαδίκτυο με ασφάλεια και αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη όταν θα θέλουμε να αναπτύξουμε κατάλληλε στρατηγικέ προστασία. Ω προ τον τόπο με τον οποίο εκμεταλλεύονται τα παιδιά οι δράστε, ε, είτε online είτε offline, μέσω ε, πορνεία ή πορνογραφία, δεν μπορούμε συνήθω ε, να βρούμε τι γίνεται με την ίδια εκμετάλλευση. Κάθε παιδί θα πρέπει να θεωρείται θύμα ε, και μπορεί να είναι ε, θύμα γιατί μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο οποιοδήποτε. Δυστυχώς τα νομικά πλαίσια είναι αρκετά αδύναμα και γι' αυτό ακριβώς ε, ζητούμε να βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κατοικοποίηση και να δούμε και τα προβλήματα στη ρίζα τους. Να μην εστιάσουμε μόνο στις εκδηλώσεις των προβλημάτων. Χρειαζόμαστε μια συστημική προσέγγιση με κοινέ δράσεις από πολλαπλούς ενδιαφερόμενους σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένες και στεναρής νομοθεσίας, διαδικασίες που τιμωρούν την εκμετάλλευση και την κακοποίηση των παιδιών και όπως ακούσαμε σήμερα ε, πολλά από τα αιτήματα είναι για περισσότερες και αυστηρότερες ποινές. Ε, Πολλές φορές ε, τα εγκλήματα αφορούν διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, αγόρια ή κορίτσια και οι δράστες εκμεταλλεύονται κάθε φορά τις αδυναμίες τους. Θα πρέπει λίγο περισσότερο να εξετάσουμε την πλευρά της ζήτησης. Επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και την παιδεία ως τρόπο εξοικείωσης των παιδιών και γνώσης και επίσης να δημιουργήσουμε μια νέα γενεά για όλους αυτούς που ε, σχετίζονται και ε, είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης λόγω πορνείας. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν ε, προγράμματα και ανάπτυξη συγκεκριμένων στρατηγικών. Βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τη βούληση των παιδιών, τις δυνατότητές τους, ε, την επινοιωτικότητά τους και το γεγονός ότι ε, μπορούν και τα ίδια τα παιδιά να μας βοηθήσουν να καταπολεμήσουμε τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση. Θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη ισορροπία μεταξύ αντιμετώπισης σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης και από την άλλη την προσωπική τους ανάπτυξη ε, και θα πρέπει να ε, βασίζονται τα παιδιά περισσότερο στην ε, βοήθεια από άλλα παιδιά και στην αυτοβοήθεια. Χρειαζόμαστε μηχανισμούς και υπηρεσίες και όλες οι προσπάθειες για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης θα πρέπει να διαθέτουν τις περισσότερες, τις καλύτερες βάσεις δεδομένων συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων από τα ίδια τα παιδιά. Θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί καταγγελίες διαθέσιμοι στα παιδιά, να είναι ασφαλείς αυτοί οι μηχανισμοί ή να είναι καλά διαφημισμένοι και να υπάρχει εύκολη πρόσβαση από πλευράς παιδιών. Επίσης υπάρχει ανάγκη για διεθνή συνεργασία, αλλά υπάρχει και ανάγκη για διασχίδεση μεταξύ δικαστικών και αστυνομικών υπηρεσιών και επίσης ε, τον τομέα της υγείας ε, της ευημερία των παιδιών και της παιδείας που ορισμένες φορές είναι οι φορείς στους οποίους αναφέρονται τα περιστατικά από τα παιδιά. Ε, και φυσικά χρειαζόμαστε και πιο αγαστή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών επειδή υπάρχει και ο σεξουαλικός τουρισμός, η συνεργασία θα πρέπει να εκτείνεται πέραν των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχουμε χώρες προς Ανατολάς και προς Δυσμάς, διότι πολλές φορές ε, ε, η σεξουαλική κακοποίηση ξεκινάει από τις αναπτυσσόμενες χώρες και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τα προβλήματα στις χώρες αυτές. Ορισμένες φορές ε, οι αυστηρότεροι νόμοι μπορεί να οδηγήσουν τους δράστες σε άλλες ε, χώρες με χαλαρότερη νομοθεσία. Με χαρά διαπιστώνουμε ότι η πρόταση οδηγίας ε, προσπαθεί να ακολουθήσει μια συνολική ε, προσέγγιση για τη σεξουαλική ε, εκμετάλλευση και την ενδιαφέρει και η προστασία και η πρόληψη. Έχουμε δώσει διεξοδικά σχόλια για την οδηγία και τα έχουμε αφήσει στην είσοδο γιατί μπορείτε να τα δείτε. Να επαναλάβω συντομία κάποια σημεία τα οποία ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τη UNICEF. Εμείς ε, προτείνουμε η ορολογία που χρησιμοποιείται για τα εγκλήματα να συνάδει με την ε, δήλωση για του, του Παγκοσμίου Συνεδρίου για τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση των παιδιών, να μην χρησιμοποιούμε όρους όπως παιδική προνογραφία, παιδική πορνεία και παιδικό σεξουαλικό τουρισμός. Προτείνουμε να δώσουμε έμφαση στην εκμετάλλευση των παιδιών στην πορνογραφία, στην πορνεία και στον σεξουαλικό τουρισμό. Επίσης μας ενδιαφέρει η αναφορά του σχεδίου οδηγίας για το συμφέρον των παιδιών ε, και το να ακούγεται και η άποψη των παιδιών για ε, την προστασία των παιδιών. Μας ενδιαφέρουν επίσης άλλες βασικές πτυχές, ε, την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, το δικαίωμα στην έλλειψη διακρίσεων και στην επιβίωση και στη σωστή ανάπτυξη των παιδιών. Όταν μιλάμε τώρα για την ηλικία συγκατάθεσης μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, θα πρέπει να λάβουμε και τα κατάλληλα μέτρα. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί αυτορύθμισης για να ε, προλάβουμε ε, τη σεξουαλική εκμετάλλευση αλλά και το σεξουαλικό τουρισμό. Ακούσαμε πολλά σήμερα για τις ποινές και θέλουμε οι ποινές να είναι ισοδύναμε με εξίσου σοβαρά ε, εγκλήματα και να εφαρμόζονται και καταλήγολος. ε, πολλές φορές διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν οι κατάλληλες ποινές αλλά δεν εφαρμόζονται όπως πρέπει. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν και ανθρώπινοι αλλά και οικονομικοί πόροι για την σωστή εφαρμογή των νόμων. Μας ανησυχεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει ε, αρκετή προστασία στα παιδιά τα οποία είναι θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Όλα τα παιδιά θύματα θα πρέπει να προστατεύονται από δίωξη όχι μόνο για εγκλήματα που σχετίζονται με πορνεία αλλά και με οτιδήποτε άλλο ώστε να μην ε, ε, να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά δεν θα πέσουν και πάλι θύματα. Επίσης χαιρετίζουμε και θα μια νέα αιτιολογική έκθεση ε, σκέψη συγγνώμη στο κείμενο που θα καλεί όλα τα κράτη-μέλη που δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση για την ε, παιδική πορνογραφία και την παιδική εκμετάλλευση να την κυρώσουν το συντομότερο δυνατόν. Υιοθετώντα την οδηγία θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα βήμα ε, προ τη σωστή κατεύθυνση και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι βασίζεται στι βέλτιστε πρακτικέ ε, στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει η Μέρη Μπανώτη, η οποία υπήρξε επιμακρών ευρωβουλευτής αλλά σήμερα εκπροσωπεί το Διεθνές Κέντρο ε, Αγνοωμένων και Παιδιών που είναι θύματα εκμετάλλευση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα δεν είμαι εδώ ως πρώην μέλος, αλλά ως εκπρόσωπος του Διεθνούς Κέντρου για τα παιδιά που έχουν ε, πέσει θύματα εκμετάλλευσης και που έχουν εξαφανιστεί. Ε, είμαι εδώ δηλαδή ως ε, αντιπρόεδρος του ε, κέντρου αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ήδη δημιουργήσει την δήλωση του τη διακήρυξη του Δουβλίνου που αφορά την αντιμετώπιση της εκμετάλλευσης στο διαδίκτυο των παιδιών. Αυτό είναι το σχέδιο του Δουβλίνου, όπω το ονομάζουμε. Ω οργανισμό είμαστε ιδιαίτερω ικανοποιημένοι που βλέπουμε ότι πολλέ από τι τότε συστάσει μα αντικατοπτρίζονται σε αυτή την οδηγία. Οπότε σύντομα θα τι διατρέξω. Θα διατρέξω τα θέματα τα οποία μας ικανοποιούν. Συμφωνούμε απόλυτα με τον ορισμό του παιδιού και δεν θεωρούμε ότι οποιοδήποτε παιδί κάτω από τα 18 είναι σε θέση να, συγκαταθε... να δώσει τη συγκατάθεσή του για την οποιαδήποτε εκμετάλλευση. Επίσης συμφωνούμε ότι ο ορισμός της παιδικής πορνογραφίας ορίζεται και ότι αυτός ο ορισμός συμπεριλαμβάνει και το ίντερνετ και τους υπολογιστές και τη σχετική ε, ορολογία. Επίσης ε, υπάρχουν ρήτρε στον ε, ποινικό κώδικα που μιλά για ποινικοποίηση της ε, ενσυνείδητης κατοχής παιδικής πορνογραφίας με σκοπό να διαβιβαστεί, να μεταδοθεί και να, ή να χρησιμοποιείται για κατέβασμα ιστοσελίδων από το ίντερνετ και εικόνων. Οι ποινικέ ε, ε, κυρώσει ε, θα πρέπει να είναι αυστηρέ και θα πρέπει να έχουν να κάνουν και με την αντιμετώπιση του κατά πόσο το παιδί συμμετείχε σε όλο αυτό ή όχι. Οι διατάξει που αφορούν το grooming ποινικοποιούν την προσέλκυση στο ίντερνετ. Τα αδικήματα αυτά τιμωρούνται και τα άτομα που βρίσκονται. Και το θέμα είναι να ποινικοποιηθεί, να τιμωρηθεί ο άνθρωπο αυτό που βρίσκεται πίσω από αυτό το έγκλημα, χωρί να πρέπει να ε, περιμένουμε για να γίνει πρώτα το έγκλημα και να τον τιμωρήσουμε εκ των υστέρων. Επίση, ε, οι κοινωνικέ ε, υπηρεσίε, οι καθηγητέ, τα όργανα επιβολή του νόμου, οι επαγγελματίε τη της ε, τεχνολογίες της πληροφορίας και άλλοι φορείς ε, πρέπει να παίξουν τον ε, ρόλο που τους αναλογεί εδώ. Επίσης, η θυματοποίηση των παιδιών από την, από την παιδική, λόγω παιδικής πορνογραφίας αναφέρεται στην οδηγία και το καλωσορίζουμε. Επίσης, οργανωμένο έγκλημα. Ε, συμπεριλαμβάνεται εδώ στην έκθεση Επίσης η διασυνοριακή μετακίνηση σημαίνει ότι ε, ζούμε σε έναν κόσμο που δεν ισχύουν πλέον οι παλαιοί κανόνες. Τα παιδιά γίνονται εμπορεύματα που, είναι, ε, που διατίθενται προς πώληση. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το στυλιτεύσουμε σε οποιαδήποτε χώρα και αν συμβαίνει. Και φυσικά συμφωνούμε ε, απόλυτα με το πώς αναφέρεται στην οδηγία, γιατί ήταν και δική μας άποψη. Ένα θέμα που δεν άκουσα όμως να συζητείτε σήμερα και το οποίο θεωρούμε ότι είναι πολύ καινοτόμο, είναι η ανησυχία που υπάρχει μεταξύ, του συνδέσμου μεταξύ παιδικής πορνογραφίας και οικονομικών συστημάτων που από κοινού με τους, ε, ε, με τους, με τους υπόλοιπους, ε, με τα εθνικά κέντρα εξαφανισμένων παιδιών, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα. Πολλοί από όσου είστε εδώ έχετε, μας έχετε επισκεφθεί στην Ουάσιγκτον και προσπαθήσαμε να δούμε κατά πόσο υπάρχει οικονομικό οικονομικός σύνδεσμος με την παιδική πορνογραφία. Και σε αυτό μας βοηθούν και οι βιομηχανίες και ο ιδιωτικός τομέας. 34 εταιρείε μα έχουν βοηθήσει στην προσπάθεια αυτή, συμπεριλαμβανομένων ε, μεγάλων ε, εταιριών πιστικών καρτών, τραπεζικών, ε, τραπεζών, εταιρείε πληρωμή τρίτων μερών κλπ. Καθώ επίση προσπαθούμε να συνεργαστούμε και με τι αρχέ επιβολή του, του, του, του νόμο ώστε να μπορέσουμε να κλείσουμε αυτούς τους λογαριασμούς και να, ε, να τιμωρήσουμε αυτούς τους ε, παράνομες επιχειρήσεις. Υπάρχει 50% πτώση στις ε, μεμονωμένες ιστοσελίδες που αφορούν την παιδική πορνογραφία, αυτά από τα δεδομένα που έχουμε από τη ΣΥΠΑ και πολλές από αυτές τις εμπορικές ιστοσελίδες χρησιμοποιούν μη παραδοσιακές μεθόδους πληρωμών και ε, βάζουν περιορισμού στις ε, βίζες που έχουν εκδοθεί ε, στις ΕΙΠΑ. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την, αυτές τις πληροφορίες ως συμβουλευτικό όργανο για, την, για το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Κέντρο που ασχολείται με το θέμα. Το Διεθνές Κέντρο επίσης ε, προσπαθεί να ενισχύσει την εργασία που γίνεται στην ε, Οικονομική Συμμαχία με μέσω προσπαθειών για δημιουργία περιφερειακών δικτύων και στη Λατινική Αμερική και στον ε, Ειρηνικό. Ε, υποστηρίζουμε ε, το φιλτράρισμα και το μπλοκάρισμα των ιστοσελίδων. Παρ' όλα αυτά, κατανοούμε ότι αυτό δεν είναι πανάκια για τα πάντα, για να αποτραπούν ε, οι περιπτώσει παιδικής ε, πορνογραφίας. Δεν μπλοκάρεται δηλαδή το υλικό στην πηγή του. δεν εξασφαλίζεται ότι το υλικό που έχει διαγραφεί δεν θα ξαναεμφανιστεί σε κάποια άλλη ιστοσελίδα. I should point out, um, it's not on my script, which I understand you have already received, that... Μιλώντας εξ ονομάτως του Διεθνούς Κέντρου, ξέρω ότι η Αμερικανική νομοθεσία διαφέρει σε κάποιες περιπτώσεις από την Ευρωπαϊκή. Η ελευθερία της έκφρασης ε, στην ΕΙΠΑ είναι ένας, ε, καταλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της νομοθεσίας. Ο βασικός μας απότερος στόχος είναι να μπορέσουμε να σταματήσουμε την επαναδιανομή κάποιων εικόνων, την παραγωγή τους και τώρα συνεργαζόμαστε με την βιομηχανία για να γίνει αυτό. Με τη Microsoft, ας πούμε. Είμαστε σε στενή συνεργασία. Για να κλείσω, είναι σαφέ ότι δεν υπάρχει ένα, μία λύση εύκολη και άμεση που να μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στη ρίζα του. Η προσβασιμότητα του ίντερνετ και οι διάφορες τεχνολογίες online έχουν δώσει στους εγκληματίες τα μέσα για να μπορούν να κατεβάζουν, να βλέπουν, να, δια... να... να ανταλλάσσουν τέτοιο υλικό που βασίζεται σε πορνογραφικές εικόνες. Που θα πρέπει να πω, Πρόεδρε, ότι... Όταν κάναμε το 2002 στο Δουβλίνο την ε, διάσκεψή μας, κανένας από εμά και κανένας από την πλειοψηφία των πολιτών που δεν εμπλέκονται σε όλη αυτή την, ε, ε, ε, τη διαδικασία κατάλαβε τι εννοούσαμε. Θεωρούσαμε ότι αυτό ήταν απλώς έτσι ένα ίσονο σημασίας θέμα και χαίρομαι που πολλοί από τους οργανωτές που παρίστανται σήμερα εδώ και συμπεριλαμβάνω και την Eurojust επίσης δεν γνώριζαν την έκταση του προβλήματος τότε. Οπότε χαίρομαι που τώρα έχουμε καλύτερη εικόνα και πιο ρεαλιστική εικόνα του τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο δίκτυο είναι σημαντική. Είναι αυτό που πρέπει να αντιμετωπίσουν. Είναι ένα έγκλημα κατά των παιδιών. Και χαίρομαι και είμαι ευγνώμων που μας δώσετε την ευκαιρία να είμαστε εδώ σήμερα για να βοηθήσουμε και εμείς τις συζητήσεις σας. Ευχαριστώ. Eh, ευχαριστώ πολύ. Είναι 6.30. Νομίζω ότι μπορούμε να διακόψουμε και να συνεχίσουμε αύριο το πρωί στις 9 το πρωί. Μας περιμένει πολύ ενδιαφέρουσα και μακρά δουλειά το πρωί. Έχουμε πολλούς ε, ομιλητές, πολλές οργανώσεις αύριο το πρωί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και στους διερμηνείς.